Λάμπερ.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 Welcome to our session, this, or our sessions in this week. Καλημέρα σας ε, στη συνεδρίασή μας. Ε, σας χαιρετίζω όλους. Ε, καλή σας μέρα. Και θεωρώ ότι δεν έχετε αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Τότε στο σημείο 2 θα ήθελα να σας ε, επισημάνω σε ανακοινώσει του Πρόεδρου ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο η έκθεση Τόγια δεν θα εξεταστεί. Βραχυπρόθεσμη ήταν η ενημέρωση ε, για την ακύρωση και την αντικαθιστούμε το σημείο αυτό με το 12 ε, για την Ένωση για τη Μεσόγειο της κυρίας Τζαβέλα. ελπίζω λοιπόν να ενημερωθήκατε όλοι έγκαιρα. Τώρα, όσον αφορά την ε, ψηφοφορία που έλαβε χώρα την Πέμπτη, ή για την Πέμπτη, που θα, με συγχωρείτε χώρα την Πέμπτη, παραμένει σε 9.30, μάλιστα παραμένει 9.30, εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Αύριο λοιπόν, 9.30 ώρα, ε, και σήμερα το 5, όπω είπαμε, ε, διαγράφεται και αντικαθίσταται από το 12. Συμφωνείτε όλοι? Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 3 της ε, ημερήσιας ε, διάταξης, το ίντερνετ ε, των πραγμάτων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπάτια Ικούτσετ. Πολύ ωραία. Σας θυμάμαι από την επίσκεψη που κάναμε στην Ισπανία. Ε, καλωσορίσατε λοιπόν θερμά και θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε καλέσει και δύο εμπειρογνώμονες ε, που θα τοποθετηθούν και αυτοί και θα σας ήμουν ευγνώμων αν ε, μπορούσαμε το χρόνο μας να τον εκμεταλλευτούμε με το σωστό τρόπο. Επίσης ε, να πω ο κύριος Κρίς και ο κύριος Βόμποντα είναι οι δύο εμπειρογνώμονες τους οποίους θα τους ακούσουμε μετά την εισηγήθεια στην οποία και δίνω το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω που καλέσαμε αυτούς τους εμπειρογνώμονες για τόσο επίκαιρα θέματα και αρκετά περίπλοκο. Θα χαρώ ιδιαίτερα να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις τους και οι υποδείξεις τους για την έκθεση αυτή. Πάνω από 40 χρόνια πέρασαν από την πρώτη εμφάνιση του ίντερνετ ε, και είχαμε μια συνεχή διαλειπτή εξέλιξη και έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο άτομα που είναι συνδεδεμένα Ξεκίνησα το 1990 στις Ηνωμένε Πολιτείε και ε, είναι το λέω και πιο δημοφιλές το μέσο και έχουμε έτσι αυτή την επαφή ανάμεσα σε άτομα και πράγματα μπορούμε να πούμε και μέσω την τεχνολογία δε ε, εξεύρεσης μέσω ραδιοσυχνότητας είναι έχουμε ένα τσίπ, μια αντένα και το τσίπ είναι ε, ένα μίκρον ε, και μπορούμε να έχουμε, μάλλον ένα χιλιαστό συγγνώμη, και χωρίς καλώδιο μπορούμε να έχουμε μεταβίβαση στοιχείων ε, και έτσι θα αντικαταστήσει τη σημαντική τεχνολογία και σε σχέση με ό,τι χρησιμοποιείται σήμερα. Βλέπουμε ότι το τσίπ δεν χρειάζεται κάποια επαφή όπως είναι με τις μαγνητικές αυτές συχνότητες ούτε χρειάζεται κώδικο με γραμμές και επίση μπορεί να συμπεριλάβει πάρα πολλές πληροφορίες ε, Σχετικά δε με τις εφαρμογές του ίντερνετ ε, στα επίκαιρα θέματα, ήδη χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές και διάφορες εφαρμογές. Να σας πω ότι στα αυτοκίνητα αυτά τα chips ε, αμέσως μπορούν να μας δείξουν ας πούμε την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου και στο ε, τρόφιμα μπορούμε να δούμε την ε, υγιεινή των τροφίμων και μια καλύτερη ανιχνευσιμότητα. Στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουν αυτά τα τσίπς και στα εθνικά τους διαβατήρια. Για το μέλλον δε, η ανείχνευση με ραδιοσυχνότητα με ένα κατάλληλο πρωτόκολλο ίντερνετ θα έχουμε έτσι ένα τεράστιο δίκτυο και το παράδειγμα ας πούμε των ψυγείων που με κατάλληλη ε, ρύθμιση θα μπορούν να μας λένε ποια είναι ε, τα προϊόντα που έχουν λήξει στο εσωτερικό τους. Αυτό θα πρέπει να δούμε τώρα βέβαια και τα θετικά και τα αρνητικά στη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Και στις 18 Ιουνίου του 2009 η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα δράσης νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Και θα πρέπει να σας πω επίσης ότι συμμερίζομαι τις γενικές γραμμές. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει προσεκτικά να εξετάσουμε εάν το νομοθετικό σημερινό πλαίσιο είναι το κατάλληλο μπροστά στην ε, μελλοντική εξέλιξη του συστήματος ή μήπω θα ε, πρέπει να έχουμε και άλλες ε, έρευνες για πτυχές σημαντικές, κυρίως όσες επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών και την ιδιωτική τους σφαίρα ζωής. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε τι γίνεται με τα ρημαγνητικά κύματα στις επιπτώσεις στην υγεία, την ανακύκλωση αυτών των chips στην ιδιωτική σφαίρα ζωής ακριβώς των πολιτών, το δικαίωμα του να, είναι, να μπορεί κανείς να διακόψει λειτουργία των chips και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων για να έχουμε μια επιτυχή εξέλιξη θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες σε αυτό το προϊόν και θα πρέπει να έχουμε ένα νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο που να προστατεύει τον καταναλωτή, των Ευρωπαίων όπως επίσης και τις επενδύσεις ιδιωτικέ και τις δημοσίες στον τομέα αυτό. Έχουμε έτσι μια μεγάλη ευκαιρία οικονομική και δυνατότητες πολλές και βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, της κατανάλωσης ενέργειας με καλύτερες, καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια ηγετική θέση σε αυτή την αγορά, μπορούμε να το κάνουμε, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα δραστήρια σε αυτόν τον τομέα, προωθώντας την έρευνα και τα πλατικά σχέδια. Ζητώ από την Επιτροπή αυτά τα σχέδια, του, ε, τα προγράμματα του 7ου προγράμματος πλαισίου, να τα υποστηρίξει και οικονομικά και επίσης για την καινοτομία, για την ανταγωνιστικότητα, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό αυτό τομέα. Όλα αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ίντερνετ και θα πρέπει να τα δούμε και στα πλαίσια της καθημερινής ζωής και την οργάνωση ας πούμε των δημοσίων μεταφορών, το ξεφορτώμα σκουπιδιών, να δούμε ποιες είναι οι αιστείες ρήπανσης, τι γίνεται με την κυκλοφορία και θα πρέπει να δούμε και την πράσινη τεχνομεκαλύτερη με καλύτερη χρησιμοποίηση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζοντας όμως το πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο μια κατάλληλη ρύθμιση νομοθετική και γι' αυτό χαίρομαι για την πρόθεση της Επιτροπής μέσα στο 2010 να παρουσιάσει μια ανακοίνωση για την ε, προστασία των ε, ιδιωτικών στοιχείων, προσωπικών στοιχείων και επίσης θα πρέπει να είμαστε υπέρ μια σωστή εφαρμογή των ρυθμίσεων που ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υιοθετηθεί και την παρουσίαση πριν από το τέλος του 2010 ενός χρονοδιαγράμματος για τους προσανατολισμούς που σε κοινοτικό συνεργή κλίμακα θέλουν να προτείνουν για την ασφάλεια της ε, έρευνας μέσω ραδιοκυμάτων. Επίσης χρειάζεται μια διεθνή συμφωνία πάνω σε αυτό. Το ίντερνετ των πραγμάτων είναι μια πραγματικότητα, μια δυνατότητα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και να έχουμε μια ηγετική θέση στην αγορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο επιτυχώς θα πρέπει όλοι να έχουν εμπιστοσύνη, όλοι οι χρήστε. Και αυτό εάν προστατεύσουμε το σύνολο των δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε και τη συνέπειες που μπορούν να υπάρξουν αρνητικά στους χρήστες. Να δούμε πώς θα προσέξουν το θέμα. Ακούω τώρα δε τις υποδείξεις στο θέμα αυτό και σας ευχαριστώ. Ich äh, darf als ersten dem Herrn Σας ευχαριστώ. Ο Δόκτωρ Κρίς έχει το λόγο. Sie Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω. Ανδρέας Κρίς είναι το όνομά μου και είμαι από τον αρμόδιο φορέα από μια όργανωση ευρωπαϊκή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων. Το 2002 ιδρυθήκαμε και συστάθηκε ο φορέας μας και εμείς δημοσιεύουμε κάθε δύο εβδομάδες μια σχετική επιστολή από το 2003 στα γερμανικά από το 2006. Εδώ πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο αφορά τα βιβλία, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικές συσκευές, ε, διατροφή, ε, είδη ρουχισμού κλπ. Είναι το ολοκληρωμένο περίπλοκο σύστημα. Τα συστήματα λοιπόν αυτά είναι συστήματα FEE e, τα οποία βοηθούν ε, στο να μπορεί κανείς ε, να παρακολουθήσει την κυκλοφορία. Κατά τα άλλα, ε, πρόκειται για τις εφής e μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας και για εφή e συστήματα δικτύων. Ε, τώρα, όσον αφορά το ίντερνετ των πραγμάτων, ε, δεν συνδέεται με το ίντερνετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Μπορεί να πρόκειται για τοπικές εφαρμογές, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα κλειστό δίκτυο, ε, το οποίο κατ' ουσίαν δεν έχει σχέση με το διαδίκτυο που γνωρίζουμε. Πρόκειται κατ' ουσίαν για ένα κλειστό δίκτυο. Και αυτό είναι μία θα είναι μία από τις πρώτες εξελίξεις αυτού του διαδικτύου των πραγμάτων πραγμάτων ε, θα έχει συγκεκριμένες εφαρμογές οι οποίες ε, θα ε, έρθουν, θα συνδεθούν με το ίντερνετ, το διαδίκτυο το οποίο γνωρίζουμε σήμερα. Όσον αφορά λοιπόν το διαδίκτυο των πραγμάτων, αυτό μπορεί να ενταχθεί ε, στα συστήματα που υπάρχουν σήμερα, ε, σε management και σε συστήματα για ε, μεταφορές και ούτω καθεξής. Ένα παράδειγμα για ευφυή συστήματα μεταφορών, έχω εδώ ένα παράδειγμα που μπορώ να σας δείξω, βλέπουμε ότι στην οθόνη μπορείτε να δείτε ότι ο σχεδιασμός ταξιδιού ε, μπορεί να γίνει μέσα από συστήματα που συνδέονται με το ίντερνετ, να ανακαλέσει κανείς πληροφορίες. Παράλληλα όμως ε, οι δημόσιες μεταφορές ε, έχουν συστήματα τα οποία ενημερώνουν, παραδείγματος χάρη, για το πότε θα έρθει το επόμενο λεωφορείο. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες τα συστήματα ασφαλείας για τους δρόμους να τα εφαρμόσει κανείς καλύτερα με την έννοια ότι σε επικίνδυνα σημεία μπορούν να συγκεντρωθούν πληροφορίες για αυτά τα σημεία και εφόσον υπάρχει ανάκληση των στοιχείων να μπορεί κανείς να δει μπροστά του ε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Κατόπιν, εκείνο που παίζει ρόλο είναι σε επόμενη φάση να συνδέσει κανείς τα αυτοκίνητα μεταξύ τους έτσι ώστε να ε, προκύπτουν και χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση στους αυτοκινητόδρομου. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο έχουμε μία σειρά διαφορετικών εφαρμογών και συστημάτων τα οποία αντιδρούν, ε, διάφορα αντικείμενα ε, τα οποία και αυτά συνδέονται μεταξύ τους, είτε το σύστημα πλοήγησης των αυτοκινήτων, είτε τα αυτοκίνητα τα οποία συνδέονται. Έχουμε λοιπόν μία σειρά διαφορετικών συστημάτων ε, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και με τον τρόπο αυτό προκύπτει μία βελτίωση της υποδομής των μεταφορών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το ίντερνετ των πραγμάτων. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά άλλα όπως τα συστήματα ενέργειας που σα ανέφερα και προηγουμένω. Τώρα, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, έχουμε λοιπόν μία σειρά σημαντικών πραγμάτων, ε, πράγματα τα οποία ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν για το ίντερνετ των πραγμάτων. Το πρώτο είναι ότι το σύστημα αυτό από τη φύση του πρέπει να συγκεντρώσει πάρα πολλά δεδομένα τα οποία πρέπει και να αξιολογήσει έτσι ώστε από αυτά τα δεδομένα να δίνει άλλες πληροφορίες τις οποίες θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να εργάζεται αποτελεσματικότερα. Άρα δηλαδή έχουμε ε, μία πληθώρα πληροφοριών που συγκεντρώνονται και την χάνουν επεξεργασίες και εδώ πρόκειται για διαφορετικά συστήματα. Δεν πρόκειται για ένα μεγάλο, αλλά για μικρά, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έχουμε δεδομένα που έχουν σχέση με άτομα, αφορούν ε, σημεία, χώρο, αφορούν την επικοινωνία, αλλά υπάρχουν και ευαίσθητα δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη ε, δεδομένα που αφορούν στην υγεία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν τίθεται το εξή ερώτημα. Ποια είναι η νομική βάση για τέτοιου είδους συστήματα. Στην προστασία των δεδομένων υπάρχουν τρεις δυνατότητες ε, για να προκύψει μια νομική βάση δεδομένων. Το ένα είναι μια ε, νομοθετική εντολή. Το δεύτερο είναι μια ε, συμφωνία, μια σύμβαση ανάμεσα στο άτομο και σε εκείνον που επεξεργάζεται δεδομένα και το τρίτο είναι η συνένεση, η ε, συγκατάθεση του ε, εν λόγω ανθρώπου για τον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να ε, συγκεντρωθούν δεδομένα, να υπάρξει αυτό το σύστημα και τι το εξή ερώτημα. Ποιο είναι εκείνο που θα χειρίζεται το σύστημα, άρα δηλαδή χρειαζόμαστε μια πολύ καλή βάση για το ποιε ακριβώ ε, πληροφορίε ε, πρέπει να την χάνουν επεξεργασίε και πάνω σε ποια νομική βάση. Διότι λόγω του όγκου των δεδομένων είναι δυνατόν να υπάρξουν βέβαια και πάρα πολλέ καταχρήσει. Φτάνουμε λοιπόν στο ερώτημα Ποιο επεξεργάζεται τα δεδομένα και ποια είναι η αρμόδια αρχή για την επεξεργασία των δεδομένων. Όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων, αυτό που παίζει ρόλο είναι ε, να καθορίσουμε τις σχέσεις ανάμεσα σε εκείνον που επεξεργάται δεδομένα και στην υπηρεσία που δίνει την εντολή για την επεξεργασία των δεδομένων κάθε φορά ο άνθρωπος για τον οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί. Τι είδου δεδομένα συγκεντρώνονται για το άτομό του, πώς μεταφέρονται αυτά και ούτω καθεξής. Και για να γίνει αυτό πρέπει κανείς να γνωρίζει την αρμόδια υπηρεσία. Επίσης, ε, ποιο θα δώσει περαιτέρω τις πληροφορίες και πώς μπορεί ο άνθρωπος να διαφυλάξει τα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερη ε, προσοχή ε, για ότι επειδή τα συστήματα κάπου την χάνουν επεξεργασία ε, στο παρασκήνιο, να ξέρει κανεί ε, περί τίνο πρόκειται. Για μεμονωμένα λοιπόν άτομα χρειαζόμαστε τη δυνατότητα ελέγχου πάνω στα συστήματα να μπορεί κανείς ε, να αποφασίσει μόνος του κατά πόσον θέλει να συμμετέχει σε ένα σύστημα ή όχι. Και επίσης να έχει κανείς τη δυνατότητα να αποκοπεί από ένα σύστημα να έχει κανείς το δικαίωμα ε, να αποσυνδεθεί από τα τσίπ. Επιγόντως λοιπόν ε, χρειαζόμαστε τη συρρήκνωση ή την περιχαράκωση των δεδομένων που συγκεντρώνονται ε, και τον ε, τρόπο με τον οποίο την χάνουν επεξεργασίας. Χρειαζόμαστε επίσης πολύ καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων περί προστασίας δεδομένων. Χρειαζόμαστε ενισχυμένους φορείς επιτήρησης οι οποίοι να έχουν και το επαρκές προσωπικό, για να μπορούν να λειτουργήσουν και χρειαζόμαστε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια καλύτερη εκπαίδευση για την συγκέντρωση δεδομένων. Αυτό πρέπει να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Και εδώ λοιπόν, κατά την άποψή μου, καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, οργανώσει την εναρμόνιση των δεδομένων και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλες χώρες για να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας ε, δεδομένων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, παγκόσμια κριτήρια για ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και εδώ όπως σας λέω ε, προκύπτει ένα ιδιαίτερο καθήκον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνοψίζοντας να πω ότι ε, πάρα πολλά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας ε, μέσα από το ίντερνετ των πραγμάτων. Οι άνθρωποι με μονομένα άτομα ε, πρέπει να έχουν τον έλεγχο πάνω σε αυτό το ίντερνετ των πραγμάτων, να υπάρχει προστασία, να περιοριστούν οι στόχοι, τα δεδομένα από κοινού με τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτή. Η δική μου οργάνωση, ο δικός μου φορέας, συνεργάζεται ε, στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε από το ίντερνετ των πραγμάτων να καταλήξουμε στο ίντερνετ των ανθρώπων και θέλουμε να υπολογίζουμε στην προστασία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μίλος Σβόμποντα, ο οποίος επίσης είναι εμπειρογνώμων.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 ε, για το θέμα της επιστοποίησης, ε, όπως λοιπόν ε, είδαμε σήμερα ή αν θέλετε όλο και περισσότερο είναι σημαντικό το να γνωρίζουμε ότι οι μηχανές θα επικοινωνούν όλο και περισσότερο μεταξύ τους. Έχουμε περίπου 5 δις ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ταυτοποιηθούν ε, και έχουμε περίπου 50 δις ευφύ e συστήματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και επικοινωνούν. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι η επικοινωνία αυτή ε, πρέπει να διασφαλίζεται και κατόπιν τούτου είναι σημαντικό να μπορεί κανείς ε, να έχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη μορφή επικοινωνίας ε, και επίσης και να διασφαλίζεται και η αξιοπιστία. Τώρα, τι είναι απαραίτητο? Μισό λεπτό, αλλά ε, εδώ αυτό που βλέπετε είναι άλλη παρουσίαση, λάθος παρουσίαση, καμία σχέση με τη δική μου. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε σε τελική ανάλυση είναι η ασφάλεια και για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια χρειαζόμαστε την εμπιστευτικότητα, ε, την ταυτότητα, ε, την ε, απόδειξη και επίσης και την πιστοποίηση. Και εδώ θα ήθελα να σας επισημάνω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Σήμερα όταν θέλει κανείς να πιστοποιήσει κάτι, αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι ε, πιστοποιεί κανείς κάποιον, αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για το πρωτότυπο. Και για να μπορεί κανείς να αποδείξει το πρωτότυπο, ε, χρειάζεται την ε, πιστοποίηση. Αυτή λοιπόν είναι η πρόκληση, όλο και περισσότερο, γιατί αν θέλουμε να επικοινωνούν 50 δις συστήματα μεταξύ τους, πρέπει να είναι και απόλυτα σαφές ε, με ποιες μηχανές επικοινωνούν μεταξύ τους τα συστήματα. Υπάρχει λοιπόν μία μέθοδος η οποία είναι γνωστή στους ε, περισσότερους. Δηλαδή, σήμερα ε, μπορώ ε, να πάρουμε ένα chip και εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα στα λογιστικά είναι να μπορούμε να πιστοποιήσουμε το προϊόν. Το θέμα είναι το εξής. Μπορούμε να πιστοποιήσουμε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Γι' αυτό λοιπόν ε, σήμερα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ένα τσίπ. Σε τελική ανάλυση υπάρχει ένας ε, αναγνώστης ε, που ρωτάει το τσίπ τον αριθμό, το τσίπ δείχνει τον αριθμό και έτσι λοιπόν μπορούμε να πιστοποιήσουμε το περί τίνος προϊόντος πρόκειται. Όσον αφορά το θέμα της πιστοποίησης ε, είναι πολύ εύκολο κοντά να υπάρχει ένας δεύτερος αναγνώστης και να ε, αντιγράψει αυτόν τον αριθμό και αργότερα επειδή ένα τσίπ είναι πολύ εύκολο να περιγραφεί, πολύ εύκολα η πληροφορία αυτή μπορεί να μεταβιβαστεί σε ένα άλλο τσίπ και με τον τρόπο αυτό ε, τα φέρνει κανείς ε, να ε, κατασκευάσει πάρα πολλούς κλόνους, κλωνοποιημένα chip. Σήμερα λοιπόν με τον τρόπο αυτό ένα chip δεν μπορεί να ε, ερευνηθεί κατά πόσο είναι πράγματι το αυθεντικό, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όπως σας είπα, στη τελική ανάλυση ένα chip δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία τράπεζα δεδομένων και πολύ εύκολα μπορεί να περιγραφεί. Όταν λοιπόν γνωρίζει κανείς την πιστοποίηση, τότε ε, πολύ εύκολα μπορεί να προχωρήσει. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει η κρυπτογράφηση. Και νομίζω όλοι ε, γνωρίζετε σήμερα πώς μπορείτε να πιστοποιηθείτε ε, σε σχέση με τον προσωπικό υπολογιστή. Ο υπολογιστής χρειάζεται έναν αριθμό και μέσα από τον αριθμό αυτό μπορείτε να πιστοποιηθείτε απέναντι στον υπολογιστή σας. Αυτό λοιπόν αποκαλείται συμμετρική ταυτοποίηση ή συμμετρική κρυπτογραφία. Νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε ότι στην πρακτική η δυσκολία έγκυται στο εξής. Σήμερα, εάν κατορθώσουμε ή αν επιθυμούμε να ε, πιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι ο αναγνώστης πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το μυστικό. Αυτό λοιπόν είναι μια ιδανική επίθεση για τον hacker, ο οποίος θα προσπαθήσει ε, στα χέρια του να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες και με τον τρόπο αυτό, μηχανές ανάγνωσης εννοούμε, και με τον τρόπο αυτό ε, να μεταφέρει τις πληροφορίες σε ένα άλλο τσίπ. Στην πρακτική λοιπόν η συμμετρική προσέγγιση για την κρυπτογραφία αφενός είναι ιδιαίτερα ασφαλής, από την άλλη πλευρά βέβαια όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικά για τη τελική ανάλυση ε, κάθε ε, μηχανή ανάγνωσης ε, πρέπει να προστατεύεται, τα μυστικά επίσης να προστατεύονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν υπάρχουν πολλές μηχανές ανάγνωσης, αυτό πρακτικά δεν είναι εφαρμόσιμο. Και τώρα θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω κάτι που δεν είναι εύκολο ε, για τον απλό άνθρωπο. Υπάρχει μια ασύμετρη προσέγγιση της ε, κρυπτογραφίας η οποία προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα. Και όλα αυτά λειτουργούν με τέτοιο τρόπο. Στον προσωπικό σας υπολογιστή δεν έχετε κανένα μυστικό, αλλά έχετε ένα δημόσιο κλειδί, μια κλίδα και με βάση αυτή την δημόσια κλίδα μπορείτε να κάνετε μία ερώτηση στο chip. Μία οποιαδήποτε ερώτηση. Μία ερώτηση που το chip δεν μπορεί να απαντήσει. Μία ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί μόνο εφόσον έχει κανείς στην κατοχή του ένα μυστικό. Αυτό λοιπόν το chip έχει το μυστικό ε, υπάρχει η κόκκινη κλίδα και με βάση την κόκκινη κλίδα μπορεί κανείς να δώσει την απάντηση. Αν δεν υπάρχει το μυστικό, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα και η απάντηση λοιπόν μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ε, το chip ακούει την απάντηση και μπορεί πολύ εύκολα να κάνει την ε, εξακρίβωση. Μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν όμως ε, ακούσει την απάντηση, μπορεί πολύ εύκολα να εξακριβώσει κατά πόσο πρόκειται για τη σωστή απάντηση. Ε, τώρα, το τεράστιο πλεονέκτημα της ασύμετρης κρυπτογραφίας έγκυται στο ότι στη μηχανή ανάγνωσης δεν χρειαζόσαστε κάτι το απόρριτο, ένα μυστικό. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ναι, δεν μπορείτε να ακούσετε την επικοινωνία, αυτό όμως δεν σας βοηθάει και πάρα πολύ και τούτο διότι κατ' ουσίαν κάνετε μόνο μία ερώτηση και ως απάντηση δεν παίρνετε το μυστικό αλλά το συμπέρασμα που συνάγεται από το μυστικό. Έχετε λοιπόν στη διάθεσή σας μια γκάμα ερωτήσεων, απίθμενη γκάμα ερωτήσεων και έτσι λοιπόν ο, την επόμενη φορά η συσκευή ανάγνωσης θα υποβάλει νέα ερώτηση. Για να καταλάβετε ας πούμε πόσες ερωτήσεις μπορεί κανείς να, υποβάλει. Υπάρχουν περίπου 260, 260 δις ερωτήσεις απίθμενος ε, όγκος ερωτήσεων όπως σας είπα, ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα αφενός να μην χρειαζόσαστε μυστικά στον προσωπικό υπολογιστή και αφετέρου η επικοινωνία δεν μπορεί να ε, παρακολουθηθεί και εφόσον ακόμα και παρακολουθηθεί την επόμενη φορά εσείς θα κάνετε άλλη ερώτηση. Αυτή είναι η περίφημα ασύμετρη προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διαμορφώσετε σήμερα τα τσίπ. Ξέρετε γιατί. Γιατί στο μέλλον όλοι θα έχουμε ε, μια τέτοια συσκευή ανάγνωσης και θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο χωρίς μυστικά να μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσον ένα τσίπ είναι πρωτότυπο ή όχι. Και αυτό μάλιστα μπορούμε να το πράξουμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και η ασφάλεια έγκυται στο ότι σε αυτό το chip περιλαμβάνεται αυτό το μυστικό κλειδί. Και σήμερα, αν προσπαθήσετε να αποκτήσετε αυτό το μυστικό κλειδί του chip, αυτό θα σας κοστίσει 500.000 ευρώ. Εκείνο όμως που επιτυγχάνουμε είναι το εξής δεν μπορείτε να ε, διαρρήξετε την υποδομή, μόνο ένα κλειδί μπορείτε να διαρρήξετε και όλα τα άλλα παραμένουν ασφαλή. Σε σχέση με την συμμετρική κρυπτογραφία, αν κανείς ε, διαρρήξει το κλειδί μια φορά, τότε έχει διαρρήξει κατ' ουσίαν όλη την υποδομή. Αυτή λοιπόν είναι η προσέγγιση η οποία κατά την άποψή μας στο μέλλον θα προσφέρει την πιστοποίηση με απλό τρόπο και προσιτό οικονομικά. Τώρα τίθεται το εξής ερώτημα. Υπάρχει ένα τέτοιο τσίπ. Διατίθεται. Σήμερα υπάρχει τέτοιο τσίπ ως πρωτότυπο. Μπορεί κανείς να αποδείξει ότι όλα αυτά λειτουργούν. Όμως ε, δυστυχώς αυτά τα chip δεν ε, παράγονται εν σειρά. Αυτό που υπάρχει είναι ότι όποιο σήμερα κάνει πιστοποίηση λέει ότι όσον αφορά στην ε, αποδειξιμότητα συσσαγωγικά οι περισσότεροι άνθρωποι παρετούνται αυτής, γιατί είναι πιο ακριβή. Ως εκ τούτου εμείς ε, απευθύνουμε έκκληση στην Επιτροπή και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η ασφάλεια μπορεί να υπάρχει μόνο εφόσον έχουμε και τους απαραίτητους κανόνες και αν γνωρίζετε ποια είναι η τεχνολογία εκείνη που ε, διατίθεται τότε υπάρχει και η νομοθετική δυνατότητα όλα αυτά να τα ε, ενσωματώσει κανείς σε κατευθυντήριες γραμμές. Και με τον τρόπο αυτό στο μέλλον όλοι οι πολίτες θα μπορούν να αποδείξουν ή να διαπιστώσουν μόνοι τους κατά πόσο ένα φαρμακευτικό προϊόν είναι πρωτότυπο ή όχι. Ε, αυτή λοιπόν η παράκληση από εμάς προς εσάς να ε, συντάξει την οδηγία έχοντας κατά νου όλα αυτά που είπαμε σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που δώσατε. Ε, συνάδελφοι τώρα έχουν ζητήσει το λόγο. Ο συνάδελφος κύριος Λάμπερς είναι ο πρώτος. Ε, ο σκιώδης ηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο αμέσω, γιατί θα πρέπει να φύγω για μια άλλη συνεδρίαση επιτροπή ε, ευθύ αμέσω. Οπότε ε, ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή και από εσά γι' αυτό. Καταρχά, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ ακριβή σύνταξη της έκθεσης και για τα ουσιαστικά στοιχεία που περιλαμβάνει. Συμμεριζόμαστε εδώ την άποψη ότι η τεχνολογία RFID και το ίντερνετ για τα πράγματα δίνουν δυνατότητες τεχνολογικές για να πετύχουμε μια οικονομία περισσότερο αποδοτική από άποψη ενέργειας και πόρων, ιδίως στον τομέα των, ε, της προμήθειας που χρειαζόμαστε, αλλά και στον χώρο του RDF. Εδώ μπορούμε να ενισχύσουμε το δυναμικό των κοινωνιών, να χρησιμοποιήσουμε ένα καλύτερο τεχνολογικό δυναμικό. Ελπίζουμε ότι θα εμπιστευτούν αυτά τα συστήματα βέβαια και οι πολίτε μας. Διότι, όπως τα είπε η συγγήτρια, είναι συστήματα σιωπηλά, αρκετά διακριτικά. Βεβαίω, κάποιο μπορεί πάντοτε να φοβάται ότι τον παρακολουθεί ο μεγάλο αδερφό, ο Big Brother. Όμω, Αυτά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως προσχήματα για να μην εφαρμόσουμε την τεχνολογία, αλλά ως ε, ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε για να επιταχύνουμε την εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων. Εάν λοιπόν κάνουμε τροπολογίες στην έκθεση αυτή, θα πρέπει να είναι χαμηλών τόνων, περιορισμένες, ήδη δηλώθηκε ότι χρειαζόμαστε διαλειτουργικότητα, αλλά νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα ήδη αυτό ισχύει σε έναν βαθμό. Τώρα, αν θέλουμε να επιταχύνουμε την ε, θέτηση των ε, τεχνολογικών λύσεων, το ένα ζήτημα είναι η προστασία του ιδιωτικού βίου και το άλλο τα πρότυπα. Προκειμένου να μπορέσουν διάφοροι φορεί να χρησιμοποιήσουν τα τεχνολογικά αυτά μέσα. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν, στηρίζουμε την έκθεση και αν έχουμε τελικά προτάσει, να είναι περισσότερο επί τη μορφή και όχι επί τη ουσία. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Ε, ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια γι' αυτό για την ανακοίνωση της Επιτροπής και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ευχαριστήσω την Οσογήτρια για αυτή την πολύ καλή της εργασία στην προετοιμασία της έκθεσης. Να θίξω όμως και ορισμένα βασικά προβλήματα. Μας μίλησαν οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί για το ίντερνετ των πραγμάτων. Δεν είναι καθαρά τεχνολογικό και μόνο φαινόμενο σύνδεσης ανάμεσα στα πράγματα και στο ίντερνετ. Το ίντερνετ των πραγμάτων, το λέει και Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, πρόκειται εδώ για ένα νέο είδος. Και η Επιτροπή αναφέρεται σε αυτό το φαινόμενο σαν κάτι που θα αλλάξει την ε, προσωπική μας κοινωνική μας ζωή στο μέλλον. Θα επηρεάσει λοιπόν τα πράγματα πάρα πολύ πολιτιστικά. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Μιλάει για κοινωνικές και πολιτιστικές λοιπόν σημαντικότητες επιπτώσεις, αλλά αναφέρεται σε δύο πτυχές, την τεχνολογική και σε αξίες όπως η ιδιωτική σφαίρα ζωής που θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν. Με την ε, παρουσίαση αυτών των τροπολογιών θα ήθελα να πω τι λείπει για τις πολιτιστικές κοινωνικές συνέπειες και στην ζωή της κοινωνίας μας στο σύνολό της. Επίσης, κάτι ακόμα που λείπει και και και Επιτροπής και στην έκθεση βλέπουμε ιδιαίτερα αισιόδοξου τόνους. Βέβαια, πρόκειται για κάτι το καινούριο, μια καινοτομία πολύ σημαντική τεχνολογική, πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό για τις μεταφορές, για την υγεία, για διάφορες πτυχές, αλλά να σκεφτούμε και τις αρνητικές πτυχές μετά από την εισαγωγή της νέας αυτής τεχνολογίας θα πρέπει από τώρα να τα εξετάσουμε για να τα προλάβουμε. Όταν μιλάμε για κοινωνικά, πολιτιστικά και τις συνέπειες αυτών, για να επιστρέψω στο πρώτο σημείο, Έχουμε να κάνουμε εδώ με πολλές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ανάμεσα στις περιφέρειες ε, για την ε, πρόσβαση στο ψηφιακό τομέα, στα κομπιούτερ, ε, στους υπολογιστές, στο ίντερνετ. Όλα αυτά δείχνουν μια διαφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνειδητοποίηση των ατόμων και στην ικανότητα των ατόμων ε, που είναι ηλικιωμένα, που είναι λιγότερο μορφωμένα για την πρόσβαση σε όλα αυτά. Και κατά κάποιο τρόπο είναι κάπως ε, απομονωμένα, αποκλεισμένα από το ίντερνετ. Είναι ένας κόσμος πάρα πολύ μπερδεμένο και δυστυχώς με όλα αυτά τα καινούργια οι διαφορές θα γιγαντωθούν. Αυτά λοιπόν θα πρέπει ιδιαίτερα να τα συλλογιστούμε για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε κατάλληλα ώστε οι κοινωνικές αυτές ομάδες και οι περιφέρειες οι οποίες αποκλείονται να μπορέσουν να συμμετάσχουν τελικά για να μην γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο το χάσμα για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, γιατί το ίντερνετ των πραγμάτων σε ορισμένες περιφέρειες, σε περιοχές θα ισχύσει τάχιστα, ενώ αλλού δεν θα υπάρξει ή θα απορριφθεί. Γι' αυτό θα πρέπει αυτά τα κοινωνικά να τα λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας. Και κάτι ακόμα για την μόρφωση, για την κατάρτιση, την εκπαίδευση της γνώσης. Δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό. Νομίζω ότι ο κ. Δικαστήλιο αναφέρεται στην έκθεσή του για το ίντερνετ. Θα πρέπει να υπολογίσουμε την πτυχή γνώση πάνω σε αυτό και στην έκθεση στην οποία μιλάμε. Θα έχω λοιπόν και από δική μου πλευρά θα παρουσιάσω, θα καταθέσω μια τροπολογία. Και ακόμα ένα σημείο. Δεν μιλάμε αρκετά για τα λάθη, για τις καταχρήσεις. Αν έχουμε ένα πολύ μπερδεμένο δίκτυο δύσκολο, περίπλοκο. Κάθε λάθος ε, στο δίκτυο αυτό θα έχει απρόβλητες ε, επιρροές ε, κοινωνικές. Είναι ένα πολύ διαδεδομένο δίκτυο και δεν πρόκειται για κάτι το... δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο ισχνό. Ε, υπάρχουν λοιπόν καταχρήσεις πέρα από τα λάθη. Με το ίντερνετ έχουμε ε, ευρύτερες καταχρήσεις πάνω σε αυτό και θα πρέπει να το συλλογιστούμε, παραλαμβάνω ιδιαίτερα όσον αφορά το ίντερνετ. Θα πρέπει με την Επιτροπή να καταρτήσουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα δράσης που να δείξει αυτή τη νέα τεχνολογία για, την, ε, το ίντερνετ των πραγμάτων. Η νέα αυτή τεχνολογία αποτελεί μια πραγματική αλλαγή για την κοινωνία μας. Στην ε, ανακοίνωση και στην έκθεση αναφέρεται η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας ε, ζωής. Θα πρέπει να το διευρύνουμε αυτό και με τις βασικές αξίες, όχι μόνο ιδιωτική σφαίρα ζωής, ότι μπορεί να παραβιαστεί θα πρέπει να αναλογιστούμε και την καλή λειτουργία αυτού του δικτύου και να σεβαστούμε αξίες όπως χάρη τη διαφάνεια, την ελευθερία, έκφρασης ελευθερία, λόγου, το να μπορεί κανείς να αποχωρήσει από αυτό το δίκτυο. Άρα λοιπόν ναι για την προστασία της δικής σφαίρας ζωής αλλά προστασία και των υπολείπων αξιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαψνόσκι, ε, σκιώδης συγητής. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτό το άριστο πραγματικά κείμενο. Νομίζω ότι έρχεται στην κατάλληλη στιγμή τώρα που πρέπει να δείξουμε πώς έχει κατάσταση με ένα φαινόμενο που το βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας με τις νέες τεχνολογίες και με τις νέες αυτές εξελίξεις όπως αναφέρει και ο συνάδελφος. Όπως το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό ξεκινώντας να λάβουμε υπόψη μας νομοθεσία που απαιτείται για να προστατεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην περιπλέξουμε τα πράγματα ακόμα περισσότερο νομικά. γιατί η τεχνολογία στην περίπτωση αυτή θα είναι αρνητική αντί ενώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα θετική. Να προσέξουμε λοιπόν ώστε να μην έχουμε αρνητικέ επιπτώσεις ε, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων που είχαμε πει λίγο πριν και θεωρώ ότι χρειάζεται να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, το είπαν και οι συνάδελφοι, για να μην ε, εμφανιστούν όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες. Ο καθένας θα πρέπει να το προσέξει, να δούμε πώς ε, θα υποφεληθούμε από τις θετικές πτυχές και όχι να μας επιβαρύνουν οι αρνητικές. Μετά από όλες αυτές τις παρατηρήσεις ε, θα τις παρουσιάσουμε και γραπτός ε, και θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε νομοθετικό επίπεδο, να μην ε, παρεμποδίσουν την ε, ανάπτυξη της τεχνολογίας και να μην, πει να μην σημειωθεί επιστοδρόμηση. Άρα λοιπόν θετικό αυτό. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια για την άριστη, τον εισηγητή για την άριστη εργασία του. Ο κύριος Λέντσου, ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον, ε, την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο, συντάσσοντας την έκθεση αυτή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο προεγνώμονες που ήρθαν μαζί μα σήμερα, διότι νομίζω με τις ε, παρουσιάσεις τους κατάφεραν να απαντήσουν σε καποιε απορίε μα και σε ερωτήματα που σκοπεύαμε ούτως ή άλλως να θέσουμε σήμερα. Το ίντερνετ των πραγμάτων είναι σίγουρα μια αναγκαία έννοια που θα αξιοποιηθεί στον κόσμο του αύριο. Και αυτό γιατί θα μας παράσχει όλα τα τεχνολογικά μέσα που διατίθενται για την ανθρωπότητα και που θα της είναι χρήσιμα. Ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη και πραγματικά να κατανοήσουμε το εξή. Εάν θέλουμε να παρακολουθήσουμε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό γύρω μα, στον υπόλοιπο κόσμο δηλαδή, θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό το ίντερνετ όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί και πάλι θα μείνουμε πίσω. Όπω λοιπόν είπε και η συγγήτρια και ο κύριο Κύ μα ε, θύμισε, υπάρχει και αρνητικό αντίκτυπο ε, λόγω τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογικών μέσων. Ο κύριος Σφόποντα μας υποσχέθηκε ότι η τεχνολογία RFID δεν απειλεί σε καμία περίπτωση το παραμικρό. Ωστόσο, πιστεύω ότι όπως έχουμε δει να συμβαίνει επανειλημμένος, οποιαδήποτε τεχνολογική λύση θετείται με σκοπό να μας προστατεύσει, μπορεί να είναι και αντικείμενο παραβιάσεων ή ε, από αντίπαλες τεχνολογικές ε, λύσεις, ανταγωνιστικές τεχνολογικές λύσεις να υπάρξουν ε, μεγάλα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή θα πρέπει να παραμείνει σε επιφυλακή να παρακολουθεί συνεχώ αυτά τα ζητήματα, ώστε να βέβαια το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο, στην privacy όπω λέγεται, των πολιτών γίνεται σεβαστό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώ την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως πολύ σωστά το αναφέρει άλλωστε αυτό και η ανακοίνωση της Επιτροπής. Εδώ μιλάμε για τεχνολογικές λύσεις, για ενημέρωση της ε, θέσης, για ταυτοποίηση, για χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί ένα άτομο να εντοπιστεί στο χώρο, να μεταδοθούν οι δράσεις του, να παρακολουθήσουμε ολόκληρη την καθημερινή του ζωή. Εδώ λοιπόν θα έχω μια τροπολογία σε σχέση με αυτές τις συσκευές και η δική μου πρόταση θα είναι ότι πέραν του δικαιώματος να παραμένουν σιωπηλές ή να παραμένει κανείς εκτός συστήματος ή Συσκευέ αυτέ ανείχνευση θα πρέπει να ενσωματώνονται μόνο κατόπιν αίτηση του συγκεκριμένου ατόμου και όχι να είναι μέρο τη τυποποιημένη διαδικασία παραγωγή. Μιλάμε εδώ για κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, υπολογιστέ προσωπικού. Το ίντερνετ λοιπόν των πραγμάτων είναι μια έννοια χρήσιμη για το μέλλον, αλλά επειδή ξεκινάει από το παρόν και εδώ βρίσκονται οι ρίζε του, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ από σήμερα τι κάνουμε και τι σχεδιάζουμε. Το τι θα αποφασιστεί σήμερα θα επηρεάσει σοβαρά τον κανονισμό που αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ σοβαρά τι προτάσει που θα γίνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Τσουκαλά, παρακαλώ έχει το λόγο. Σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή συνεδρίαση της ΣΥΤΡΕ είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν συνδυάσουμε το συζητούμενο θέμα με το σημείο 8 που είναι το Internet Governance που θα το δούμε στη συνέχεια, καθώς επίσης και την έκθεση Ρούμπεχ για τα πνευματικά δικαιώματα. Να ευχαριστήσω θέλω την ε, κυρία εισηγήτρια για την ε, έκθεση της, καθώς και τους δύο εμπειρογνώμονες που με φώτισαν σχετικά με ζητήματα για τα οποία είχα και εγώ σκεφτεί. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι όταν φωνάξεις το διάβολο στο σπίτι σου θα χορέψεις το χορό του. Αυτή η τεχνολογία για την οποία εδώ γίνεται τόσος λόγος είναι μια τεχνολογία την οποία την ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό. Είχε άλλο όνομα, λεγόταν Ambient Intelligence και τώρα έγινε Internet of Things ενώ είναι προφανές ότι τελικά είναι ίντερνετ των ανθρώπων. Η φόβη μου δεν είναι μόνο εξαιτία του ότι αναφέρεται στην ιδιωτικότητα των πολιτών, αναφέρεται στη συγκρότηση της πολιτείας. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι δεν θέλω πάλι να αναφερθώ στον πολύ κοινότοπο πλέον Orwell, θα κάνω μια αναφορά και θα σας θυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια ένα συγγραφέας, ο David Brin, έγραψε ένα τεχνολογικό βιβλίο που λεγόταν The Tales of the Two Cities με υπότιτλο City of Control και Transparent Society. Στην προκειμένη περίπτωση, ενώ έχω ξοδέψει όλη τη ζωή μου στην τεχνολογία και την επιστήμη, παρά είμαι επιφυλακτικός σε τέτοια μείζωνα μεταβολή όχι μόνο της ατομικής ζωής των πολιτών αλλά και της διάρθρωσης των πολιτικών συστημάτων. Εξηγούμε. Παρατήρηση πρώτη. Τα πολιτεύματα αλλάζουν, η τεχνολογία μένει. Δύο. Η τεχνολογία είναι ηθική ή ανήθικη ανάλογα με τη χρήση της. Παράδειγμα, από Ανατολή ο τρόπος που η επιχειρηματική ηθική αλλάζει σύμφωνα με τις επιταγές του κράτους μέλους που παραγγέλει τις τεχνολογικές υπηρεσίες που στην Ευρώπη και στον άλλον κόσμο σηκώνουν την τρίχα όρθια. Τρίτο παράδειγμα αν θέλετε. Αναφέρατε πολύ συχνά ότι ένα πρώτο παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι η εφαρμογή εισαγωγής τσίπ στα διαβατήρια των πολιτών. Θα ήμουν πολύ ενδιαφερόμενο στη μάχη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων να μάθαινα αν σε αυτές τις χώρες που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία ο πολίτης ενημερώνεται το τι ακριβώς περιλαμβάνει το τσίπ με το οποίο εμφανίζεται στον κισέ του κάθε κράτους διαφανής και ευπρόσβλητος στις προσωπικές του πληροφορίες που κανείς δεν του λέει τι λένε. Υπό την έννοια αυτή, ενώ η έκθεση της αξιότιμης κυρίας εισηγήτριας φαίνεται να δίνει μεγάλη προσοχή στην οικονομική και τεχνολογική διάσταση της εφαρμογής του Internet of Things, μάλλον στα γρήγορα περνάει ή βιάζεται να συμμεριστεί με την έκφραση στο σημείο 2 Σημερίζεται την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδει η Επιτροπή στην ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, καθώς και την διακυβέρνηση του ίντερνετ των πραγμάτων. Προσωπικά πιστεύω, από τεχνική και νομική άποψη, η Επιτροπή δεν δίνει καμιά ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που λέμε. Το ζήτημα δεν είναι ατομικό. Το ζήτημα είναι συγκρότηση του κράτους αυτό είναι το ambient intelligence που τώρα τον λέμε Internet of Things και το οποίο θα επηρεάσει τη ζωή και την δομή των κοινωνιών των ανθρώπων. Υπό την έννοια αυτή, μολονότι γνωρίζω πολύ καλά ότι ανάγκη υπάρχει να προχωράει η τεχνολογία, δεν είμαι πρόθυμος ή έτοιμος να συμμετάσχω σε επιπόλες πράξεις που δεν θα διασφάλιζαν κάτι τι που εγώ τουλάχιστον το βλέπω να έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Gracias, eh, presidente. Κύριε Καστίγιο, ευχαριστώ πρόεδρε γρήγορα γρήγορα να ευχαριστήσω ε, την συγγήτρια για όσα μας είπε, μας παρουσίασε με πλούσιο περιεχόμενο, πολύ ευρύ, ε, τη θήγη όλες τις πτυχές ε, και εδώ η παρουσίαση βέβαια επικεντρώνεται περισσότερο και ιδιαίτερα επαγγελματικά μπορούμε να πούμε σε αυτά τα κλειδιά του ίντερνετ. Ε, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που σχετικά με την έκθεση έχουν σημασία έχουν να κάνουν και με τις τροπολογίες και με την ε, ε, εκ των υστέρων επεξεργασία, στη συνέχεια επεξεργασία της εισηγήτριας με τους ορισμούς, αλλαγές κλπ. Ίσως θα πρέπει αυτά να τα έβλεπε, θα τα πω εγώ τώρα. Καταρχήν, θα πρέπει να συνδυάσουμε την έκθεση αυτή με την σφαιρική ψηφιακή στρατηγική την οποία ακολουθούμε και στο Κοινοβούλιο και αλλού στην Ευρώπη αυτό το χρονοδιάγραμμα το ψηφιακό που θα συζητηθεί και αύριο και η Επιτροπή όπως ξέρει η γήτρια θα υποβάλει το τέλος του Απριλίου ένα χρονοδιάγραμμα ψηφιακό και επίσης εργάζεται η Ισπανική Προεδρία πάνω σε αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να το αναφέρουμε στο πλαίσιο αυτό. Είναι σημαντικό. Δεύτερο τώρα. Ειδική αναφορά στην υποστήριξη περισσότερο από την ανάγκη της πρόθεσης επιτροπής για την παρακολούθηση, την εκτίμηση αυτής της ανάγκης, επαναλαμβάνω, μιας επιπλέον εναρμόνισης του πλαισίου για το ίντερνετ των πραγμάτων. Κατά την άποψή μου σημαντικό θα ήταν να δώσουμε έμφαση γιατί το πρώτο που θα έπρεπε να ξεκινήσει είναι ότι χρειάζεται αμέσως ε, οτιδήποτε σχετικά με αυτό το εύρος, το φάσμα ε, θα πρέπει να δούμε γιατί είναι από τα σημεία κλειδιά τι όλε δέσμε στα τηλεπικοινωνιακά. Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει όλο αυτό το περιεχόμενο να μεταφερθεί όπω είναι στο framework, στο πλαίσιο αυτό και ακόμα στην ε, σε όλα αυτά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και μία αναφορά γιατί χρειάζεται να ενισχυθεί Υπάρχουν ε, οι ρυθμίσεις ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας ζωής ε, και ίσως καλύτερο θα ήταν να μιλάμε για προσαρμογή της οδηγίας, για την προσαρμογή της οδηγίας προστασίας δεδομένων στο ψηφιακό σημερινό πλαίσιο. Αυτό θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, γι' αυτό χρειάζεται να αναφερθεί μια ακόμα σκέψη για τη διατήρηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης ε, για την έρευνα και στα πλαίσια του προγραμματός πλαισίου. Θα ήθελα να πω στην ε, εισηγήτρια ότι χρειάζεται να συνεχιστούν αυτά τα πράγματα, αλλά ειδική προσπάθεια επίσης να καταβάλουμε Όσοι τα σχέδια αυτά, τεχνολογίες, επικοινωνίας κλπ. που έχουν να κάνουν με πάρα πολλούς τομείς ε, για να μην πούμε ότι έχει να κάνει σχέση, ότι έχει σχέση με όλο το φάσμα της κοινωνίας σήμερα. Ε, δεν είναι ότι λείπουν ε, μόνο πράγματα. Χρειάζεται να διπλασιαστεί η προσπάθεια και από στον ψηφιακό προγραμματισμό χρειάζεται να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να έχουμε και πολύ υψηλότερο προϋπολογισμό που να πηγαίνει σε αυτό. Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στο ότι χρειάζεται να μειωθούν όλες αυτές οι γραφειοκρατικές δυσκολίες για την πρόσβαση στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, τις δυσκολίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτό το θα πρέπει να λυθεί. Κάτι ακόμα ιδιαίτερα ενδεικτικό ήταν μια αναφορά στον ρόλο της ε, πόλης, ε, τι γίνεται εκεί, σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ε, πιστεύω ότι όπως το κάνουμε στην ψηφιακό χρονοδιάγραμμα, στην ψηφιακή ατζέντα και αλλού, αυτό, ε, αυτή η διοκτησία μπορούμε να πούμε αυτού του συνόλου, αυτού του προσανατολισμού της ανάπτυξης και η η προώθηση ψηφιακή με διάφορες ενέργειες, ε, διάφορες ρυθμίσεις, ε, όλα αυτά θα πρέπει να πάει και πέρα από τις πόλεις. Ε, στις ε, εθνικούς φορείς, στους περιφερειακούς φορείς, στους τοπικούς φορείς ε, και πόσους ασχολούνται με αυτά. Θα πρέπει να δούμε βρούμε ότι είναι μια παρότρινση που απαιτείται, χρειάζεται μια συμμετοχή από όλους τους τομείς που έχουν λόγο σε αυτό και που έχουν ευθύνη στην όλη ανάπτυξη. Χρειάζεται να συμμετάσχουν και να πλαπλασιάσουμε λοιπόν αυτή την αναφορά που αναφέρεται μόνο στον ρόλο των πολιτιών και να ευχηθώ καλή τύχη στην εισηγήτρια και ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Και Ροντή, ο επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές, καθώς και τους εμπειρογνώμονές μας. Έχοντας ακούσει όμως τους εμπειρογνώμονες, πρέπει να πω, οι παρουσιάσεις τους ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, όμως όπως το, το υπογράμμισε και ο συνάδελφος ο κύριος Τσουκαλάς, δημιουργούν και κάποιους ανησυχίες. Ας πούμε στο σημείο 8 αναφέρεται ένα σύνολο εξελίξεων για τις οποίες έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια λειτουργίας όλων αυτών των εφαρμογών. Εμένα το ερώτημά μου προς τους εμπειρογνώμονες είναι τι θα γίνει αν κάτι από αυτά ε, χαλάσει. Εάν υπάρξει ένα σύνολο βλαβών σε ένα μέρος του πλανήτη, στην Ευρώπη α πούμε. Τι θα γίνει αν είναι σε βλάβη όλα αυτά τα συστήματα. πώ θα επηρεάσουν τη λειτουργία πόλεων, κρατών που θα έχουν στηριχθεί εξ ολοκλήρου σε πράγματα εντό εισαγωγικών. Πράγματα μάλιστα εντό εισαγωγικών ευθύ. Θα έπρεπε λοιπόν σε αυτέ τι διατάξει να συμπεριληφθεί και η έννοια τη ευθύνη, ποιο είναι υπεύθυνο για όλα αυτά, προκειμένου να λειτουργούν εύρυθμα και προκειμένου να υπάρχει η ευθύνη και το υπόλογο, πρέπει να υπάρχει και η ανεχναυσιμότητα των πληροφοριών. Να υπάρχει ένα σύνολο πληροφοριών και να γνωρίζουμε από πού πηγάζουν και πού διοχετεύονται όλες αυτές οι πληροφορίες ώστε να μπορούμε με τη χρήση αυτών των τεχνολογικών μέσων και να καλύψουμε τις ανάγκες για ε, καλή διαβίωση των Ευρωπαίων, αλλά και να καταπολεμήσουμε την εξαπάτηση και τι παράνομε δραστηριότητε ενδεχομένω, καθώ και να καλύψουμε και άλλα ζητήματα όπω τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Οι ανησυχίε λοιπόν και οι ενδιασμοί αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν όλε τι ανάγκε του ιδιωτικού βίου και τη ιδιωτική σφαίρα και θα πρέπει να τι εξασφαλίσουν ε, δημόσιοι φορεί, πολιτικοί φορεί. Όχι όπω γίνεται στην Αμερική από φορεί ιδιωτικού, όπω στην ε, Καλιφόρνια που υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τα ζητήματα αυτά. Πρέπει εδώ να υπάρχει μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη ανάληψη ευθύνη για να διασφαλίσουμε το όφελο όλων μα των πολιτών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Τελευταίο ομιλητή, ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την εργασία της. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας, γιατί νομίζω ότι πηγαίνουν προς την κατεύθυνση και της ανακοίνωσή μας ε, που παρουσιάσαμε τον Ιούνιο. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Ε, εδώ δεν θα κάνω άλλα σχόλια, είπαν ορισμένα πράγματα προηγούμενο μιλητέ, αλλά θα κάνω μια διάκριση για μα σημαντική ανάμεσα στο ίντερνετ των πραγμάτων ε, και την ε, ανείχνευση μέσω ραδιοσυχνότητα, την RFID που είναι ειδική τεχνολογία. Το ίντερνετ ε, είναι των πραγμάτων καλύπτει ένα σύνολο τεχνολογιών. Οι αισθητήρε, ε, όπως και εδώ, οι σουηδικοί μετρητές που χρησιμοποιούνται παντού, είτε στα σύγχρονα πάρκιν και στις Βρυξέλλες, ε, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί είναι οι ε, προδρομοί όλων αυτών, αλλά δεν χρησιμοποιούν αυτή τη ραδιοσυχνότητα που είναι σημαντική τεχνολογία για την Ευρώπη. Είναι δύο chips ε, ανακάτοικο αντιστοιχούν και είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα αυτό, αλλά όχι όπως ε, ίντερνετ των πραγμάτων. Ε, θα πρέπει να ασκηθεί η πολιτική για τα δύο, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσά τους. Παρακαλώ προσέξτε κάτι, προσέξτε δύο πτυχές της ανακοίνωσης που μας ενδιαφέρουν πολύ. Πρώτα απ' όλα την χρήση, την αντιμετώπιση αυτού του ίντερνετ των πραγμάτων. Ε, αν τίμημα και ήταν ε, ένας στόχος ακριβώς για το σύνολο του πλανήτη και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο σημείο 8 το Intergovernmental Forum που αναφέρθηκε αρκετές φορές σήμερα το πρωί. Παρακαλώ να καταλάβετε τι γίνεται με το ίντερνετ όταν θα ενταχθούν εκεί και τα αντικείμενα της καθημερινής μας ζωής και χρειάζεται ε, το κράτος ε, παντού να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και το αποκαλούμε αυτή η διαχείριση του ίντερνετ των πραγμάτων και να μην έχουμε μια αντιπαράθεση λόγω ας πούμε και της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας πραγμάτων ε, ζωής αλλά χρειάζεται να δούμε αυτή τη διαχείριση πριν να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία, πριν να οριμάσει πλήρως ώστε να μην δώσουν απάντηση άλλοι και εμείς να βρεθούμε προτελεσμένων γεγονότων. Ποιος θα το ελέγξει αυτό το ίντερνετ, ποια θα είναι η θέση, ποια θα είναι η αρμόδια νομοθεσία, ποια θα είναι η θέση του δημοσίου είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που χρειάζεται να υποβάλουμε στους εαυτούς μας και πολλά άλλα ακόμα και τα πανεπιστήμια και η βιομηχανία μας προς το παρόν είναι ισόπαλοι με τους ξένους ε, εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει ο καθένας να παίξει το ρόλο που του αρμόζει και το ρόλο επίσης που οι πολίτες από μας περιμένουν. Ένα δεύτερο σημείο τώρα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για την προστασία των στοιχείων. Νομίζω ότι ε, το αναφέρατε πλατιά σήμερα το πρωί. Αλλά μια λεπτομέρεια στην ανακοίνωση μιλάμε στο δικαίωμα συγγής των τσίπς. Ε, το είπαν ορισμένοι υπό την ευρία έννοια ότι θα πρέπει το δικαίωμα, να έχει το δικαίωμα ο πολίτης να αποσυνδεθεί από αυτό. Πρόκειται για ένα νόημα πάνω από ένα δικαίωμα. Χρειάζεται να το διερευνήσουμε αυτό λεπτομερέστερα και να δούμε νομικά, τεχνικά τι συνεπάγεται. Δεν έχω χρόνο να αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτά, τα υπόλοιπα σημεία του προγράμματος δράσης και της ανακοίνωσης. Χαίρομαι πάντως ε, που στο διαθεσμικό διάλογο τον οποίο επιθυμούμε για αυτό το ίδιο των πραγμάτων υπάρχουν ήδη αρκετά από σήμερα που συζητήθηκαν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που αποδώσατε και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Να στραφούμε τώρα στην εισηγήτρια, εφόσον θέλετε πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες και όσους πήραν το λόγο, όπως επίσης ε, και την Επιτροπή. Στη ζήτηση αυτή ακούσαμε τη λέξη ανησυχία, κίνδυνο, κατάχρηση. Γι' αυτό ακριβώς η Επιτροπή πάνω σε αυτά που παρουσίασε, εδώ στην έκθεση εμείς με τη σειρά μας τονίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια καινούρια κατάσταση και μια καινούρια εποχή τεχνολογίας ίντερνετ που θα μπορούσε να μας διευκολύνει ιδιαίτερα, θα μπορούσε να μας βοηθήσει πολύ στη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι τρία βασικά θέματα μπορούμε να παρατηρήσουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε, όπως είπε και η Επιτροπή να προβλέψουμε από τώρα τι μπορεί να γίνει πριν να έχουμε την πλήρη τεχνολογία γιατί τότε θα είναι κάπως αργά, θα είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Πολύ σημαντικό είναι να γίνει ταυτόχρονα εργασία, συνεργασία ακριβώ με τους εμπειρογνώμονες και τους νομοθέτες ε, από νομικής πλευράς. Γιατί ίσως υπάρξουν προβλήματα λόγω των νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει να λύνονται ταυτόχρονα μέσω της τεχνολογίας της ίδιας. Δηλαδή η τεχνολογία μας προσφέρει και το θετικό και το αρνητικό και μας σωθεί σε εξέβρεση λύσεων τους θέματα που ακούσαμε εδώ. Για να δούμε τον αποκλεισμό, να δούμε τη γνώση ατόμων, ε, όλα αυτά, όχι μόνο για, την, ε, για το ίντερνετ των πραγμάτων, αλλά γενικά για το ίντερνετ. Όλα αυτά είναι σημαντικά, τα συμμερίζομαι, το θέμα της διαφάνειας, το πώς θα συνδυαστεί αυτή η πληροφορία με την όλη στρατηγική, την ψηφιακή σίγουρα και αυτό που προσπάθησε γιατί θεωρώ λογικό είναι στην έκθεση και μετά και από την ανακοίνωση Επιτροπής να την εστιάσω ισορροπημένα. Υπάρχει μια δυνατότητα που μας προσφέρεται με πολλές βελτιώσεις και χρειάζονται και εγγύησεις βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται μόνο να προβάλλουμε τον κίνδυνο. Υπάρχουν σίγουρα κίνδυνοι, αυτό που προσπαθούμε όμως είναι να δώσουμε μια ισορροπία σε αυτό, να μέσα σε όφελος και κίνδυνο. Πρέπει να εποφεληθούμε από τα πλέον εκτήματα, από τα θετικά και να προσέξουμε τους κινδύνους. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις τους και εντάξει θα χαιρόμουν να συμπεριλάβω όλες αυτές τις τροπολογίες που υποβάλλετε για να εμπλουτίσω την έκθεση και για να μπορέσω να δώσω έγκαιρα μία απάντηση σε όλα αυτά που δημιουργούν δημιουργούνται λόγω της νέας εποχής του ίντερνετ. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Απλώς να θυμίσω εδώ ότι ως τις 25 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες και ας κλείσουμε την ε, όλη συζήτηση για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Meine Damen und Herren, ich darf damit zu Tagesordnung. Κυρίε και κύριοι, Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξη, ευθύ αμέσω. και με ιδιαίτερη χαρά μου εδώ καλωσορίζω τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με διαφορετική εδώ ιδιότητα σήμερα. Ο κύριος Μπαρόν Κρέσπο λοιπόν είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει μια νέα έκθεση. Νέα έκθεση που εκπονήθηκε στα πλαίσια τη ε, Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου και Θέλουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχετε να μα πείτε γι' αυτό. Έχουμε διάφορα έγγραφα στα χέρια μα, Αλλά θα ήθελα χωρί καθυστερήσεις να σας δώσω ευθύ αμέσω το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει στα γερμανικά ο κύριος Μπαρόν. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ευρωβουλευτές, εδώ για 23 χρόνια ήμουν παρόν θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω, ξεκινώντας, το γνωρίζετε ότι αποφάσισα να μην ε, κατέβω και πάλι σε εκλογές τον Ιούνιο του 2009. Ε, διδάσκω στο Τολέδο την έδρα και επίσης με ένα μικρό ίδρυμα για την κοινωνία της πληροφορίας υπό το βελγικό δίκαιο με νεαρό κοινό γιατί νομίζω ότι η επικοινωνία είναι από τους μεγάλους άξονες τους μελλοντικού και με τον κύριο Ρος τον Υφυπουργό που είναι υπεύθυνο από Ισπανικής Προεδρίας αυτό ε, συζήτησα για το πρόβλημα αυτό και με πρότεινε, μου πρότεινε να προεδρεύσω μια ομάδα εργασίας, μιας πρωτοβουλία του συνόλου της ε, ΤΙΚ ε, βιομηχανία ενημέρωσης και δέχτηκα εγώ να προεδρεύσω, το θεώρησα ενδιαφέρον και με την εργασία αυτή με κατάλληλο συντονισμό γιατί αντιμετωπίστηκε από όλη τη βιομηχανία αυτό το θέμα έχουμε σαν αποτέλεσμα, σαν πόρισμα το κείμενο, το έγγραφο που έχετε στα χέρια σας. Θα πρέπει να σε εξηγήσω εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον που μου δημιουργήθηκε για την κοινωνία της πληροφορίας, της επικοινωνίας και παλιότερα πριν να ενταχθεί ενταχθεί η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ ήμουν στην Ισπανική κυβέρνηση, στην, υπηρεσία, στην ε, Υπουργό Μεταφορών και διαπραγματευόμαστε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ ασχολήθηκα και ε, στο ταχυδρομείο στο κέντρο της Μαδρίτης εγκατέστησα το πρώτο φαξ. Είναι προϊστορία αυτή με δεινόσαυρους και άλλα παρόμοια γιατί ναι, το 1983 είχα, ανακαλύψει το φαξ στην Ιαπωνία και ε, στο τέλεξ τότε ε, ήταν δύσκολο να γράψουν Ιαπωνέζικα, γι' αυτό ανακάλυψαν το φαξ. Και όταν έφτασα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είδα δύο παραδείγματα πώς μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας με τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής σε ορισμένε αίθουσε της Επιτροπής, όχι σαν αυτές εδώ. Ε, οι κλητήρες ε, έφερναν στον καθένα τις οδηγίες ε, και ήταν σαν κτηνοτροφικός οργανισμός εδώ πέρα. Ήταν ένα σαν παζάρι, σαν... Ε, ήταν ένα θέαμα που δεν άρμασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες οι τροπολογίες τότε το 80 θα έπρεπε να τυπωθούν. Βλέπετε πως άλλαξε λοιπόν αυτό στη ζωή μας. Προχωρήσαμε, αλλά δεν προχωρήσαμε μόνο εμείς. Αν εξετάσουμε την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία είναι στο ευρύ φάσμα οι πρωτοπόρες, χάρη σε πρωτοβουλίες ε, κρατικές. Και η Κίνα, και η Κίνα εργάζεται στο ε, πάνω σε αυτά. Να σας πω και κάτι ιστορικά, ότι υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στις ελευθερίες, στην κοινωνία και, και όπως και στη Σοβιετική Ένωση, ένα σύστημα παλιότερα που έλεγχε τις ε, τεχνικές επικοινωνίες. Χρειάζεται ορισμένα πράγματα να τα προστατεύσουμε. Και εδώ εμείς προχωρήσαμε εμείς οι Ευρωπαίοι το GSM, την κινητή τηλεφωνία, προχωρήσαμε εμεί οι Ευρωπαίοι και όταν εμφανίστηκαν τα Nokia τα τηλέφωνα, σκεφτόταν όλοι ότι ήταν Ιαπωνέζικα τα τηλέφωνα αυτά. Κανεί δεν σκεφτόταν, δεν φανταζόταν ότι ήταν Φινλανδικά. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που κέρδισαν πολλά από αυτά από τεχνικής πλευράς. Και σχετικά με την έκθεση αυτή να σας πω και ότι ξεκολουθούμε να εργαστούμε, να εργαζόμαστε. Εάν ρίξετε μια ματιά τώρα, αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς γίνεται διοικητικές σχολές διοίκησης σχετικά με τα θέματα αυτά. Θα δείτε ότι βλέπετε ε, ότι οι καλύτεροι φοιτητέ φεύγουν για την Καλιφόρνια και καταλαβαίνετε την επιτυχία των εταιριών των Αμερικανικών για να που ασχολούνται με το ίντερνετ. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Για να δούμε τώρα την αξία της έκθεσης αυτής. Ξέρετε ότι οι εκθέσεις ε, στο βιομηχανικό τομέα έχουν αυτό το προκπαταρικό αμάρτημα, όπως ο Ντάμα Σμιθ, ε, όταν πάνε τέσσερις επιχειρηματίες που πάνε και πίνουν ένα καφεδάκι, αμέσως συνομωτούν κατά των τιμών. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό. Θα δείτε διάφορες αναφορές ε, που, που κατηγορούν την αύξηση τιμών θα πρέπει να δούμε και τους πρωταγωνιστές όλων αυτών ε, είναι ανταγωνιστές ε, αδίστακτοι καμιά φορά και για πρώτη φορά ε, όλοι μαζί κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι οι μεγαλοεπιχειρηματίες αλλά και οι μικροί οι εναλλακτικοί ε, του GSM, ε, για τα ψηφιακά, οι κατασκευαστές, οι έμποροι, με τα δορυφορικά συστήματα, όλα αυτά. Το σημαντικό είναι να καταλάβει, να λάβει υπόψη της η Ευρώπη τη σημασία του ψηφιακού αυτού τομέα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω ιδιαίτερα. Θα δείτε στην έκθεση αυτή ότι υπάρχει μια σύνοψη στις πρώτες σελίδες αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά. Και εδώ βλέπετε τι αναφέρεται σχετικά. Αλλά μερικά σημεία είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Είναι μια βιομηχανία με 718 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι και που θα μπορούσε να διπλασιαστεί αυτό το ποσό σε 6 χρόνια. Ε, μπορούν επίσης να δημιουργηθούν ε, περισσότερες, πολύ περισσότερες θέσει εργασία από κάθε τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα υψηλό αριθμό απασχολούμενων που είναι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια 35 δισεκατομμύρια ευρώ οι επενδύσεις. Είναι βιομηχανία η οποία συνεισφέρει ιδιαίτερα στη μείωση της εκπομπής ε, αερίων διοξιδίου του άνθρακος ε, και αν θεωρήσουμε και ποιες είναι οι ανάγκες μεταφόρες ε, και αυτά τα βλέπει και η πληροφορική. Η βιομηχανία λοιπόν αυτή είναι πράσινη βιομηχανία σε σχέση με άλλες ε, Όλα αυτά τα πρώτα στοιχεία, τα επιχειρήματα είναι σημαντικά τώρα που συμπίπτουν τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στη δεύτερη επιτροπή Μπαρόζο τίθεται ένα θέμα για την ψηφιακή Ευρώπη και επίσης η έκθεση για την Ευρώπη 2020 ή 2020 στρατηγική να την πετύχουμε και ακόμα να θεωρούνται οι δημοσιονομικές προοπτικές. Καταλαβαίνετε και αυτό έχει τεράστια σημασία και μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα όπως την έκθεση της αναστεργασίας για το μέλλον ε, που προωθείται από τον Φελίπε Γκονθάλες ε, και την Ισπανική κυβέρνηση. Να σας ενημερώσω επίσης ότι πρόσφατα στις Βρυξέλλες πριν από δύο εβδομάδες ε, οργανώθηκε μια συνάντηση με την Ευρώπη μας στον φορέα αυτό και 14 ε, ε, λήπτες αποφάσεων ε, σχετικά με την Ευρώπη και εγώ ήμουν στο προεδρείο της όλης συζήτησης για το θέμα αυτό του μέλλοντος και χρειάστηκε να πω στους εισηγητές μας, στους εμπειρογνώμονες ότι δεν είχαν πει τίποτα για το μέλλον της ψηφιακής Ευρώπης. Βέβαια συζήτησαν για σημερινά πράγματα, τι γίνεται τώρα για την ε, αυτοκινητομηχανία, αλλά είναι κάτι που υπάρχει ήδη, αλλά δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους τη σημασία της ψηφιακής Ευρώπης και μάλιστα για το μέλλον. Ε, θα πρέπει τώρα τη στιγμή αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να παίξουν ενεργό ρόλο και θα ήθελα να ευχάσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση αυτή την ε, κυρία Δελκαστήλια, συμπατριώτησά μου. Νομίζω ότι αυτά που μας προσφέρει είναι πολύ θετικά και επίσης την κατάλληλη στιγμή πέφτουν, έρχονται αυτά. Σχετικά τώρα με το περιεχόμενο της έκθεσης, τι μπαίνει στη μέση. Χρειάζεται να δούμε πού θα παίξουμε, να δούμε, έτσι μιλάω αθλητικά τώρα, μια εσωτερική πισαγορά που να μπορέσει να λειτουργήσει το κατάλληλο γήπεδο. Εδώ προτείνονται διάφορα μέτρα. Εντάξει, τα βλέπετε και αυτά αν θέλετε εδώ στην έκθεση αυτή. Ξέρω ότι είσαστε ιδιαίτερα απασχολημένοι. Τέλος πάντων, ε, ρίξτε μια ματιά, <laughs> τουλάχιστον εδώ στο Προεδρείο. Εδώ εμφανίζονται σημαντικά στοιχεία, πρέπει να τα υπογραμμίσουμε και το είπα και ο ρόλος του ΤΙΚ στην ε, όλη αυτή η ανάπτυξη, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για το μέλλον μας και μπορείτε να το δείτε και στις περισσότερες ανταγωνιστικές οικονομίες ε, που είναι κυρίως οι βόρειες οικονομίες, ε, την ανάπτυξη της πληροφορικής του τομέα αυτού. Εκεί αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένα σημαντικό άξονα για το μέλλον για να προσφερθεί εγγύηση ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη σε ένα κόσμο όλο και πιο δύσκολο πάνω σε αυτό. Επίσης ε, το θέμα της αηφορίας Αναφέρθηκα επίσης και στη μείωση των αερίων δεξίου του άνθρακος, αλλά ε, όχι μόνο ότι αποφεύγουμε μεταφορά, μετα, αύξηση του τομέα των μεταφορών, ε, εδώ όλα αυτά, στον ειδικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, όλα αυτά είναι σημαντικά και σιγά σιγά τα συνηθίζουμε πώς θα χρησιμοποιούμε έτσι την πληροφορική και αποφεύγουμε τις μεταφορές λοιπόν και για την ενέργεια που παίζει ρόλο και όχι μόνο στα σπίτια μας για τη θερμασία και τα υπόλοιπα, αλλά και στις μεταφόρες. Ε, όλες αυτές είναι προκλήσεις λοιπόν, χρειάζεται να τα δούμε. Εδώ θα πρέπει να δούμε στον ψηφιακό τομέα την δημιουργικό χαρακτήρα όλων αυτών, η βιομηχανία, προωθεί τη φιλοσοφία της, ε, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία πολιτική και να δούμε την ανάπτυξη μιας πραγματικά ενίας αγοράς χωρίς ε, φράγματα και εμπόδια. Θα πρέπει να δούμε και την προσαρμογή δύο πραγμάτων που διαφέρουν μεταξύ τους η προστασία ε, Τη δυνατότητα παραγωγής, αναπαραγωγή στην μια μεριά, αλλά και το copyright από την άλλη. Και θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Ε, την αντιμετώπιση τους όσον αφορά αγορές ε, διαφορετικές είτε επιμέρους αγορές, να δούμε και τα συστήματα προστασίας Όλα αυτά χρειάζεται να τα λάβουμε υπόψη μα. Θα πρέπει βέβαια να είμαστε υπέρ του να υπάρχει μια ενιαία αγορά και υπέρ των καταναλωτών να είμαστε, αλλά και όσον αφορά τη δημιουργία, την επιστημονική, την καλλιτεχνική, λογοτεχνική κλπ. Η Ευρώπη είναι από του ιδιαίτερα ενεργού τομεί μα, όχι μόνο ιστορικά αλλά και στο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώ ε, θα πρέπει να θέσουμε ορισμένα ερωτηματικά επίκαιρα, πολύ σημαντικά, σε κάθε διαδικασία ψηφιοποίησης ε, της, ε, των πολιτιστικών μας στοιχείων. Τέλος πάντων, δεν θα επιστρέψω σε λεπτομέρειες, θα πρέπει να το δούμε και σε άλλα πλαίσια αυτό και να το δείτε κι εσείς, αλλά και αυτό είναι κάτι το επίκαιρο. Κάτι ακόμα θέμα εμπιστοσύνης συστήματα προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών. Το είδαμε σήμερα στην ε, έκθεση της συναδέλφου σας ε, με πολύ σημαντικά θέματα όπως το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και αυτό πολύ επίκαιρο θέμα και ήδη είναι κάτι το θετικό σαν αυτά τα δικαιώματα γιατί χάρτα, έχουμε την χάρτα των ε, θεμελιώδη δικαιωμάτων και συμπεριλαμβάνεται και η προστασία των δεδομένων. Ισχύει αυτό λοιπόν και ήμουν στη συντακτική συνέλευση το 77 στην Ισπανία και είναι από τα πιο σύγχρονα συντάγματα το ισπανικό ε, ιστορικούς λόγους, αλλά δεν μπήκε το θέμα τότε της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, γιατί δεν είχαμε την ίδια εξέλιξη σε αυτά εδώ. Είναι κάτι που εξελίχθηκε όμως, παρουσιάστηκε, εξελίχθηκε και είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται λοιπόν μια συμμετοχή και εμπιστοσύνη από όλου και επίσης η πρόσβαση στην αγορά. Εδώ λοιπόν εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου στην ε, πρώτη θητεία ήδη. Έμαθα διδάχτηκα πολλά πράγματα. Τώρα στη συνάντηση της Ντόχα τα TRIPS που είναι όλα αυτά τα θέματα τα εμπορικά που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας και την συμφωνία ΙΤΑ που είναι σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας. Όλα αυτά ε, σπρώχνουν προς αντιπαραθέσεις αλλά είναι πολύ σημαντικά έχουμε τρομερές αλλαγές και να φερθούμε και σε μια χώρα καινούρια που αλλάζει και για οικονομικούς λόγους αλλά και νομισματικούς είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Η Κίνα από τη στιγμή που μπήκε στην ΠΟΕ είναι η πρώτη αναγνώριση που ζητήσαμε από την Κίνα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τους στίξε πολλά είχε υψηλό κόστο για αυτού, δεν ήταν συνηθισμένοι, αλλά ήταν το πρώτο στοιχείο που έπρεπε να δούμε και επίσης λοιπόν για την πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να υπερασπιστούμε να ισχύουν ορισμένοι κανόνες και να του σέβονται όλοι. Και κάτι ακόμα, η μείωση του διοικητικού κόστους ε, και του φόρτου δουλειά ε, και θα πρέπει να δούμε τους ειδικού φόρους ε, στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης ε, θα πρέπει να αποφύγουμε διακρίσεις στην εσωτερική αγορά. Χρειάζεται να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας. Αυτό είναι το περιεχόμενο λοιπόν της έκθεσης. Ε, λοιπόν, οι βιομήχανοι με τους οποίους συναντήθηκα έθιξαν ε, σημαντικά θέματα και όσα μας απασχολούν στην Ευρώπη και σχεδόν όπως ε, το Κοινοβούλιο προσπάθησαν ε, να απομονώσουν τις διαφορές και να τις παρακάμψουν θα πρέπει οι υπεύθυνοι από το Δημόσιο αλλά και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, οι κυβερνήσεις στο Συμβούλιο θα πρέπει να κατανοήσουν την ε, σημαντικότητα τομέα αυτού για το μέλλον μας. Αυτά κύριε Πρόεδρε και θα ολοκληρώσω με τρεις σκέψεις, ε, όχι δικές μου προσωπικές, αλλά προέρχονται όλα αυτά από την εργασία στα πλαίσια της έκθεσης και νομίζω ότι συνδυάζονται με αυτά που ακολουθείτε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα, η κατάσταση, η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο η αναγνώριση του δικαιώματος του πολίτου στην συμμετοχή στο ευρύ φάσμα και εδώ όλα αυτά που είναι σταθετικά, νομοθετικά από διάφορες κρατήρες, ε, Φιλανδία, Εστονία, Ισπανία και επίσης ε, ο πάγο. Ε, ε, το αναγνώρισε στην το αναγνωρίζει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες χώρες. Ε, πάντως να σας πω ότι όλα αυτά αλλάζουν τα στοιχεία, τα δεδομένα δεν είναι μόνο οι βιομήχανοι που να προσπαθούν να παγιώσουν τη θέση τους και τις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές, υπηρεσίες, μεγάλη βρισδιάδρομοι, Είναι δικαίωμα όλων των πολιτών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα 500 εκατομμύρια πολίτες ε, είναι, αν είναι στη Ρουμανία, αν είναι βόρεια-βόρεια στη Φιλανδία, αν είναι στα Κανάρια νησιά ακόμα και στη νότια-νότια Κρήτη την ελληνική. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ε, όλα αυτά. Δημιουργούν ε, θέματα βέβαια και προϋπολογισμού σε ορισμένα κράτη. Έχουμε διάφορες εμπειρίες μέχρι τώρα έχει αποκτηθεί κάποια πείρα. Όλα αυτά κοστίζουν χρήματα όμως. Ε, θα πρέπει να δούμε και στην Ισπανία τι γίνεται, κάτι που θα χτιστεί πραγματικά και να δούμε τα διάφορα στοιχεία που θα βοηθήσουν για το ευρυφάσμα αυτό και να μπορέσουν οι επικοινωνίες, ε, η επικοινωνία να γίνεται και με τις πιο μακρισμένες περιοχές και επίσης ε, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί αυτό το δικαίωμα συμμετοχής. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην χάρτα δικαιωμάτων, αλλά νομίζω ότι παλιώνεται σιγά σιγά. Και ακόμα θέματα αντιφατικά, αλλά ορισμένα απασχολούν την ε, Ισπανική Προεδρία, την πνευματική ιδιοκτησία ας πούμε και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες ε, στην προσαρμογή αυτής της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε ένα πρώτο στοιχείο για τα δυτικοευρωπαϊκά συστήματα σύμφωνα με το δίκαιο από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά σχετικά με την πνευματική διακτησία και βιομηχανικά, εικόνας κλπ, ε, πλαστικές τέχνες, όλα αυτά που σιγά σιγά εξελίχθηκαν και το δικαίωμα αναπαραγωγής, τι γίνεται με αυτό, δεν έχει μόνο σχέση με τα δικαιώματα του συνδέτου εκδότη, αλλά σιγά σιγά δημιουργήθηκαν αυτά και είναι μια παράδοση από τη Βασίλισσα Άννα και μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο που διαθέτει ένα σύστημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης έχει το ίδιο σύστημα. Όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία γιατί σε σχέση με την όλη διαχείριση και όσους διαχειρίζονται όλα αυτά δεν είναι κάτι το μονοπωλιακό πέρα από όταν είναι ένα εμπόρευμα ή κάτι περισσότερο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα έχει σημασία. Όπως το γνωρίζετε, με την ανάπτυξη του ίντερνετ είχαμε τρομερές αλλαγές και ακόμα περισσότερες θα έχουμε στο μέλλον, ας πούμε στις εκδόσεις, στην παραγωγή δίσκων μουσικής ε, και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα οπτικοακουστικά και καλλιτεχνικά γενικά. Θα πρέπει να επιβεβαιωθούν τα δικαιώματα των χρηστών ε, σαν χρήστες, σαν καταναλωτές και προτείνεται μια χάρτα και μηχανισμοί αποτελεσματικοί για την προστασία των χρηστών ταυτόχρονα αλλά που να έχει σχέση με και με κάτι σημαντικό, τους πειρατές, τα εγκλήματα πληροφορικής, ε, εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες, ε, χρηματοδότηση διεθνούς τρομοκρατίας ε, και εκμετάλλευση άλλων όπως παιδική πορνογραφία. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν ε, μόνο με το δίκαιο μιας χώρας, ε, αλλά γενικότερο, τελευταίο κυρίες και κύριοι, το μέλλον των μέσων επικοινωνίας και οπτικοακουστικά και γραπτά. Δεν είναι μόνο ο Μάρντοκ που τα δημιουργεί αυτά, αλλά τα μέσα σε όλες τις χώρες μας ε, όλα αυτά έχουν και σελίδα στο ίντερνετ και πήραν μέτρα ταυτόχρονα για να μπορέσουν να επιβιώσουν ε, και το περιεχόμενό τους να γίνεται σεβαστό όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο για τη δική σας επιτροπή, αλλά η δική σας επιτροπή μπορεί να είναι μπροστάρις στον τομέα και εποφελούμε τις ευκαιρίες κύριε Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας ε, να επιβεβαιώσω ότι το να προχωρήσει κανείς στην ψηφιακή Ευρώπη είναι από τους πιο πλούσιους τομείς που εγγυώνται το μέλλον μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Im Namen des gesamten Ausschusses und äh, habe auch erste σας ευχαριστώ πολύ εξ ονόματος ε, της Επιτροπής και ε, κάποιοι συνάδελφοι έχουν αποβάλουν ερωτήσεις. Ε, η κυρία Ρέρα Μαντορέλ είναι η πρώτη. Εδώ λέει η κυρία Ντίας. Ναι, ναι, ναι, η κυρία Ρέρα Μαντορέλ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μπαρον Κάσπα που είναι εδώ. Ναι, ήταν και εδώ πρόεδρος και εγώ ήμουν πρόεδρος στην ομάδα. Να σας, δώσω, να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας με το συντονισμό αυτής της σημαντικής έκθεσης για τη βιομηχανία, για τεχνολογία, επικοινωνίες και το είπατε πολύ σωστά ότι για ακόμη μια φορά δείχνει το σημείο κλειδί αυτό τον ΤΙΚ ε, στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ε, και όπως το δείχνει εδώ η όλα αυτά παίζουν σημασία για χαμηλότερες εκπομπές αερίων διοξιδίου του άνθρακος με καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ε, στους Ευρωπαίους, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να προετοιμάσει τα εργατικά χέρια στην Ευρώπη για τις εργασίες αυτές και καλύτερη κατάσταση στην Ευρώπη ανταγωνιστικά σε μια παγκόσμια αγορά. Και επίσης όλες αυτές τις δυνατότητες για να τις εκμεταλλευτούμε χρειάζεται να υποφεληθούμε από τη συντονισμένη προσπάθεια των δημοσίων φορέων και των οικονομικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου. Στη μελέτη του κυρίου Μπαρόν, νομίζω ότι η μελέτη αυτή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Για πρώτη φορά έχουμε να κάνουμε με ένα τομέα που έχει μία και μόνο φωνή, ενιαία, δείχνει αυτό που μας ενώνει και όχι αυτό που μας χωρίζει. Επίσης είναι μια ανάσα δροσερού αέρα σε αυτή τη συζήτηση για μια δροσερή πνοή για τις τηλεπικοινωνίες όπου κανονικά ισχύει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε πρώην ε, μονοπωλιακούς παράγοντες, χρήστες, διοικητικούς, ε, ε, τη κινητή επικοινωνία, δίκτυα και κατόχους δικαιωμάτων και όλα αυτά. Τώρα, πέρα από τις συγκεκριμένες από την Ισπανική Προεδρία και που σίγουρα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και στην Καστήλιο σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αυτό το ψηφιακό που θα ψηφιστεί αύριο. Θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή τη νέα δυναμική που είχαμε και ελπίζω και άλλες προεδρίες και άλλοι φορείς και ειδικότερα εδώ το Κοινοβούλιο να διατηρήσουν και να ενισχύσουν. Έχουμε προκλήσεις τρομερές για αυτά τα ψηφιακά για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα επικοινωνία με καινοτόμες λύσεις και ενωμένο τομέας και όχι διαιρεμένο. Θα ήθελα να ρωτήσω και το πρώτο. Νομίζετε ότι τα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στη συνεργασία ανάμεσα στους στα ενεργά μέλη στον τομέα αυτό και ακόμα κάτι σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά. Από ό,τι φαίνεται μόνο το 7% των συναλλαγών είναι διαμεθοριακές. Τι γίνεται με αυτή τη λειτουργία που δεν είναι τόσο θετική με αυτή τη δραστηριότητα. Τίποτα άλλο περισσότερο και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Μπαρόν γνωρίζει ότι είναι το σπίτι του εδώ. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του και ευχόμαστε να συνεχίσουμε μαζί του τη συνεργασία και στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Κύριε ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ δεν θα ρωτήσω τίποτα, αλλά θα εκφράσω μερικές σκέψεις και απόψεις μου. Για τον κύριο Μπαρό να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα εδώ να τονίσω ότι πραγματικά εκείνος δείχνεται ευαίσθητος όπως και φορέας του για αυτή την εξέλιξη και την επανάσταση, την ψηφιακή και όλα τα στοιχεία, όλους τους παράγοντες που έχουν να κάνουν με την επανάσταση αυτή, ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί η Ευρώπη από αυτή την επανάσταση, ό,τι γίνεται περισσότερο και καλύτερο για την ευμάρεια της κοινωνίας ευχόμαστε και για την ανάπτυξη, για την απασχόληση και για όλες τις κοινωνικές πτυχές που καθορίζονται από την ανάπτυξη αυτή. Οι περισσότερες λοιπόν θέσεις απασχόλησης, ο τομέας αυτός έχει ηγετική θέση και δεν χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο. Δείχνει όμως και την ευαισθησία της Ισπανικής Προεδρίας που ιδιαίτερα υποστηρίζει την ανάπτυξη της έκθεσης αυτής και να πω κάτι. Εμφανίζεται επίσης ε, στα διάφορα όργανα και στους διάφορους φορείς και τομείς ε, ότι υπάρχει μια κάποια συνεργασία προς την αυτή κατεύθυνση για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η Ευρώπη όσο γίνεται περισσότερο να αποφελήθει από τις δυνατότητες αυτής της ψηφιακής εποχής. Σχετικά με όσα είπε η συνάδελφος ε, Ριέρα Μαδουρέλα, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα ενταχθούν, πώς θα υπάρξει μια διευκόλυση για τα μέσα για να προχωρήσουμε στην την ε, ευχόμενη κατάσταση για μια πλήρη απασχόληση ώστε να έχει ο κόσμος γνώσεις για να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή για να γνωριστούν και τα δικαιώματα όλα αυτά όλες αυτές οι ανάγκες ε, χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθεί ο τομέας, ο ψηφιακός με την κατάλληλη από μας παρακολούθηση και όταν ε, τα πράγματα είναι σαφή συγκεκριμένα και οριστικά, φάνονται και τα προβλήματα αν υπάρχουν διαφορετικές πριοπτικές ε, ε, και διαφορετικοί στόχοι από κάθε πλευρά στα πλαίσια αυτής της νέας ε, ψηφιακής δέσμης. Εδώ όλα αυτά να πω ότι βοήθησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ισορροπημένη θέση, ένα πλαίσιο που να έχουμε λογικά διαφορετικές απόψεις ε, όταν απαιτείται και ακόμα σε αρκετά θέματα στα πλαίσια αυτά, στα χρονοδιαγράμματα ψηφιακά και του Κοινοβουλίου που αύριο ψηφίζεται και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τέλος του Απριλίου όπως επίσης στη Γρανάδα της Ισπανικής Προεδρίας. Θα, όλα αυτά θα πάνε και στο Συμβούλιο μετά και θα πει και το Συμβούλιο αρκετά. Όταν όλα αυτά λοιπόν προχωρούν και μπαίνουν στα πλαίσια ειδικών ρυθμίσεων εδώ και εκεί σε ειδικέ αποφάσεις ε, θα δούμε, θα διαπιστώσουμε αυτές τις διαφορές, αλλά δεν θα πρέπει να μας φοβίζει αυτό. Ποιο είναι το σημαντικό σε αυτή την παρουσίαση που μας έκανε ο κύριος Μπαρό, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Όλα αυτά αποδεικνύουν και πάλι ότι υπάρχει ένας συνδυασμό ένας κοινό ορίζοντας προς τον οποίο ατενίζουμε όλοι μας, αυτή η διαφορετική πολιτική φόρης, αλλά και ο ιδιωτικό τομέας όλοι είναι αποφασισμένοι την ηγετική θέση της Ευρώπης στις τεχνολογίες, πληροφορίας και επικοινωνίας. Όλα αυτά όχι να μην χαθούν αλλά να ενισχυθούν. Προς την κατεύθυνση αυτή, εκεί θα πρέπει να εντάξουμε αυτή την έκθεση, όπως και το αυριανό χρονοδιάγραμμα εδώ στην Επιτροπή, με τις προτάσεις αυτές και θα τις δούμε άμεσα και συγκεκριμένα. Αυτά λοιπόν ε, νομίζουμε ότι είναι και η κατάλληλη στιγμή και το ευχόμαστε. Έχουμε ιδιαίτερη συνειδητοποίηση ότι αυτά είναι σημαντικά. Έχουμε και πολλές προτάσεις επιτάπητος και όλα αυτά νομίζουμε ότι συγκλίνουν. Ε, και γι' αυτό θα σας ευχαριστήσω και να πω ότι είμαι αισιόδοξη. Ευχαριστούμε κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομιλητή για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για την επίσης ενδιαφέρουσα έκθεση. Εδώ αναφέρεται ο σημαντικός ρόλος των ICT ως φορέα που θα προάγει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προσπάθεια μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μια από τι βασικέ προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για το μέλλον είναι η αποδοτικότητα όλων των φυσικών μας πόρων, από το νερό έως τα ορυκτά και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 η οποία θα επικεντρωθεί επίσης στη γενικότερη αποδοτικότητα των πόρων, όχι μόνο την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής και θα ήθελα να το σχολιάσετε ή δυνατόν για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, ICT, δεν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα όλων των πόρων που θα είναι τόσο σημαντικοί για την Ευρώπη στο μέλλον και ιδίω στα πλαίσια του ανταγωνισμού με τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως για πολύ αποτελεσματικά ορυκτά καύσιμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριος Οντί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυο... λόγια θα να πω στα Ισπανικά. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σε αυτό το νικό δικό σας είναι. Μαζί εργαστήκαμε στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και εσείς διατελέσατε πρόεδρος εκεί. Και τώρα να περάσω στη μετρική μου γλώσσα, πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας για τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης. Είστε ένας μεγάλος Ευρωπαίος άντρας, κύριε Κρέσκου, Απλώς θα πρέπει εδώ να ασχοληθούμε με το ψηφιακό χάσμα. Ε, μιλάμε για πολλούς στόχους αριθμητικούς, όμως στον επικράτη της Ευρώπης βλέπουμε να υπάρχει τελικά ένα χάσμα ψηφιακό. Δεν είναι ίσες οι ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, στα πλαίσια του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού ανταγωνισμού. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι έφτασε η στιγμή η κατάλληλη στιγμή για να έχουμε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά θεμάτων, για την ενέργεια, το διάστημα, αλλά σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες. Και για να μπορέσουμε να έχουμε το απαραίτητο περιεχόμενο, δηλαδή και την αποδοτικότητα. Δεν χρειάζεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών στο σύνολο των ψηφιακών υποδομών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία παρατήρηση, κυρία Τόμσον. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρόν για την παρουσία του σήμερα εδώ. Θα μιλήσω δανέζικα τώρα. Είναι προφανές ε, νομίζω ότι όλα αυτά που μας αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ε, βεβαίως όλοι πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση στις ευρυζωνικές διασυνδέσεις. Διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή ότι οι περιφέρειες χάνουν ε, όλο και περισσότερους πολίτες ε, και εκεί παρουσιάζεται ε, ύφεση, οικονομική ύφεση, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση. Οι άνθρωποι λοιπόν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και παράλληλα είναι δύσκολο να προσελκύσει κανείς νέους πολίτες περιοχές αυτές. Αυτό λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για τις περιφερειακές περιοχές. Το θέμα είναι ότι η ίση πρόσβαση πρέπει να υπάρχει για όλους, όχι μόνο στη δημοκρατία, ε, στην ιατρική. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που διαδραματίζονται μέσω ίντερνετ. Σήμερα οι ε, δάσκαλοι και οι καθηγητές, ίσως κυρίως οι μαθητές, χρησιμοποιούν περισσότερο το Google από ότι να πηγαίνουν στο σχολείο. Ε, το θέμα είναι ότι όσον αφορά την εξέλιξη δεν πρόκειται μόνο για τεχνικούς σπόρους αλλά και για ανθρώπινους σπόρους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ευρώπης δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Στη Δανία έχουμε παντού διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά το 20% των Δανών δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση του διαδικτύου. Κατά την άποψή μου λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πρόβλημα δημοκρατίας. Έχουμε την οικονομική κρίση, που άρα πολλοί άνθρωποι ε, κατέστησαν άνεργοι και τώρα λοιπόν στη Δανία διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι που έχουν γίνει άνεργοι ε, δεν έχουν και σωστή χρήση του διαδικτύου. Υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι που ε, και μαθητές που δεν έχουν διαδίκτυο και ήδη τώρα βρίσκονται σε υστέρηση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όχι μόνο να φροντίσουμε να υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση, αλλά και όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Γιατί αλλιώς πραγματικά υφίσταται τεράτιο, τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά αυτό το ε, χάσμα στην τεχνολογία. Ε, κύριε Κρέσπο, παρακαλώ να απαντήσετε. Καταρχήν, απευθύνομαι στην Τερέζα. Εσείς ε, με ρωτήσατε ε, κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των ε, θεσμών. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τους ε, θεσμούς. Είναι καθαρά δικό τους θέμα. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αυτό πράγματι είναι δικαίωμα των πολιτών. Όταν λέμε ποιοι τομείς ε, θα πρέπει να προαχθούν έτσι ώστε να σημειώνεται συνεχώς ε, πρόοδο. Ε, εγώ θέλω να πω ότι το διαδίκτυο διαδραματίζει καθοριστική σημασία ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να συνεργαστούμε, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κατόπιν αναφέρθηκε ότι μόνο το 7% των συναλλαγών είναι Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εδώ πρέπει λιγάκι να το διευκρινίσουμε. Όταν μιλάμε για μεγάλους ε, φορείς, ε, δεν θα ήθελα να κάνω διαφήμιση για κανέναν. Orange, Vodafone, Telefonica. Ήδη υπάρχει μια συνεργασία στην αγορά ε, και όλοι προσπαθούν ε, στην ε, Ευρώπη να αποκτήσουν μία θέση στην αγορά. Αν δούμε λιγάκι αυτό που προσφέρεται στο hardware και στο software, είναι πολύ δύσκολο κανείς να καταργήσει τους φραγμούς και κατόπιν εσείς μιλήσατε για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα πολύ ε, δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Ε, δεν υπάρχει δίκαιο ε, για ευρωπαϊκούς συλλόγους, για ευρωπαϊκά ιδρύματα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Ακόμα δεν έχει φτάσει αυτή η στιγμή. Όμως ε, πρέπει να είμαστε συνεπείς. Όταν θα τεθεί σε ισχύ ο χάρτης των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό θα έχει ε, πάρα πολλές συνέπειες και η πνευματική ιδιοκτησία είναι μία μορφή ιδιοκτησίας, όπου δεν πρόκειται για αντικείμενα, αλλά πρόκειται για την δημιουργικότητα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το θέμα αυτό να προαχθεί. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι επικεφαλής του Ιδρύματος Νταλή, ε, διαβίου πρόεδρος. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο Νταλή στην Ευρώπη, αλλά πάρα πολλά έργα του Νταλή έχουν παραποιηθεί. Το Ισπανικό κράτος είναι κατ' ουσίαν ε, ο κύριος ιδιοκτήτης και εγώ απλά το εκπροσωπώ. Μας κόστισε λοιπόν εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα για τις φωτογραφίες και τις εικόνες από τα έργα του Νταλή. Υπάρχει ένα πολύ καλό δίκτυο για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Υπάρχει τώρα πλέον αυτό, αλλά ε, χρειάστηκε για πάρα πολλά χρόνια να χρηματοδοτήσουμε το δίκτυο αυτό, να δαπανίσουμε πολλά χρήματα για να επιτύχουμε αυτό που κατορθώσαμε. Ε, Βεβαίω αυτό φαντάζομαι το κάνει και η Νομική Επιτροπή και η Επιτροπή Πολιτισμού, γιατί το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Η κυρία Ντεκαστήλιο το είπε και αυτή και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας ανέφερε. Η αξία αυτής της έκθεσης ε, θα μπορούσε να λειτουργήσει και είναι το ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ε, καμπανάκι συναγερμού για το μέλλον. Κοιτάξτε κύριε Καβάλιο, αν δείτε λιγάκι το πώς ε, ακριβώς διαχειριζόμαστε το νερό στη Γεωργία και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μου αλλά αφορά τις περισσότερες χώρες της ε, Μεσογείου και της Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τεχνολογίες ε, που χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση νερού είναι πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα η χρήση της ε, πληροφορικής τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι ε, καθοριστική σημασία για να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση των πόρων μας. Η τεχνολογία της επικοινωνίας ε, και της ε, τεχνολογίας είναι ο σύμμαχος του πρασινίσματος της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ θετικό. Γαλλικά, γαλλικά μιλάει. Προς τον κύριο να πω ότι αυτό που αναφέρατε για την κάλυψη όλη τη επικράτεια έχει να κάνει και με τη θέματα τη ηλικία και τη της, δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη. Όταν μίλησα για το δικαίωμα όλων των πολιτών, δικαίωμα πρόσβαση στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, εννοούσα προφανώ ότι εάν αναγνωρίζουμε αυτό το δικαίωμα, πρέπει να είμαστε και συνεπεί. Δηλαδή, Πρέπει να γίνουν και απαραίτητε επενδύσει. Προ στιγμή, το σύνολο των επενδύσεων προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, είναι σαν να γίνονται, να προβλέπονται διόδια ουσιαστικά και προκολαβία των διοδίων. Σε χώρες όπως η Ιαπωνία όμως και η Κορέα υπάρχει μια τελείως διαφορετική πολιτική. Όμω, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να αντλήσουμε κονδύλια από τον κρατικό προπολογισμό. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι, εφόσον αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα και θέλουμε να είμαστε συνεπεί, δεν θα πρέπει εν ώψη των ερχόμενων τη αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών για το ερχόμενο διάστημα και εφόσον μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχή, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε και τι επενδύσει ε, εκτός από τις ε, πιο συγκεκριμένες, τις υλικέ αυτοκινητοδρόμους, έργα, δημόσια έργα και τις άιλες και την επένδυση σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα αναγκαστικά να ταξιδεύουν. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους πολίτες να επιλέξουν και πού θέλουν να κατοικούν. Εγώ έχω εμπειρία από τη δική μου τη χώρα. Λόγω χάρη, στα 150 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη, και το γνωρίζω αυτό λόγω του Ιδρύματος, υπάρχει μια πόλη, Κουέγκα, όπου θα φτάσει σίγουρα το τρένο υψηλή ταχύτητα σε λίγους μήνες. Υπάρχουν λοιπόν πολίτε που θέλουν να εργαστούν εκεί ή άλλοι που θα ζουν στη γύρω περιοχή. Αλλά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και στο χωρί στο ασύρματο δίκτυο ίντερνετ για να μπορούν να αναπτύξουν τις βιομηχανικές τους δραστηριότητε σε εκείνη την ε, περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να αποφασίσει η βιομηχανία στη θέση μα. Η βιομηχανία όταν λαμβάνει αποφάσει και αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα μεταξύ των ε, φορέων, των βασικών φορέων της αγοράς και των αναλλακτικών, ε, έχει άλλε λύσει να προτείνει. Δεν είναι θέμα πολιτική ευθύνη. Βέβαια, από άποψη του υπολογισμού δεν είναι τώρα στιγμή να θέσουμε τέτοια ερωτήματα. Αλλά ξέρετε ότι όταν υπάρχουν δυσκολίε, η φαντασία παίρνει μεγαλύτερο ρόλο. Για την κυρία Τόμσεν, μαζί με απάντηση στον κύριο Ντί, που μίλησε για το πρόβλημα που έχει να κάνει με τις γενιές τις διάφορες. Είναι πολύ σημαντικό σαν θέμα μας ε, ανησυχεί πάντα τρομερά το τι γίνεται, πώς θα φτάσει στους πολίτες το μήνυμά μας. Γιατί βλέπουμε ότι δεν ψηφίζει ο κόσμος, δεν προσέχει αυτό που κάνουμε, αυτό που λέμε. Και περισσότεροι από τους 50% των παιδιών μας, των εγγονιών μας, ε, ε, μαθαίνουν ε, από το ίντερνετ, όχι μόνο από το facebook και το twitter. Ε, είναι δίκτυα που τα διαχειρίζονται Αμερικανοί, όπως το Google ας πούμε. Αλλά υπάρχει τηλεόραση από το ίντερνετ, η TV. Ε Γιατί να μην καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς να τα κάνουμε όλα αυτά για να δείξουμε πράγματα και στους νέους το μέλλον μας. Και ακόμα τι γίνεται με τα ψηφιακά. Και εγώ ήμουν μάρτυρας αυτής της εμπειρίας ε, και με τεχνολογία πληροφορίας. Ε, 20-30% το πολύ του πληθυσμού μας έχει κανονική πρόσβαση στο ίντερνετ. Είναι μια νέα κοινωνική ελίτ. Υπάρχει, δημιουργείται χάσμα Λοιπόν, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Πώς θα γίνει, πώς θα έχουμε μικρά terminals ε, και μέσω των δήμων, μέσω αποκεντρωμένων μονάδων ε, και να επιτρέψει στον κόσμο αυτό να έχει πρόσβαση όπως και εμείς. Ε, και εγώ παλιότερα ήμουν αναλφάβητος πληροφορικά. Εδώ με στα βρουδάκια έβαζα και τώρα χρησιμοποιώ την πληροφορική για να το ίντερνετ για να έρθω σε επαφή, να απευθυνθώ κλπ. Και στα βουνά του Κάντιθ που είναι κοντά στο Γιβραλτάρ ε, από εκεί πέρα στα βουνά πάνω ο άλλο το παιδί έχει με το συγγενή του συνομιλεί στην Ολλανδία. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία και εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να πετύχει η βιομηχανία, αλλά είναι και πολιτικές αποφάσεις για το τι θα μπορεί και πρέπει να κάνει η βιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις κυβερνήσεις, τις ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εμείς είμαστε πρωτοπόροι, θα πρέπει να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάντως που με αφήσετε, μου επιτρέψατε να αναλύσω αυτό το κείμενο και να προσφέρω και απαντήσεις που θα μπορούσα να σας βοηθήσουμε με τη σειρά σας τις εργασίες σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, για τις πληροφορίες που μας δώσατε, για την επισκεψή και ελπίζω να ξανάρθετε σύντομα. Meine ich darf äh, mit Einverständnis den nächsten Punkt aufrufen. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, αν συμφωνείτε, θα πάμε στο επόμενο θέμα, το σημείο υπεριθμών 5. Ε, το βγάλαμε από τη μερική διάταξη και προτάξαμε το σημείο υπεριθμών 12, που είναι η Ένωση για τη Μεσόγειο. Η συγγήτρια είναι η κυρία ε, Τζαβέλα, η οποία είναι ήδη εδώ και ως εκ τούτου της δίνω ευθύ αμέσω το λόγο και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, να τις αφιερώσουν την προσοχή τους. Παρακαλώ κυρία Τζαβέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις που έχω κάνει ε, για την Ευρωμεσογειακή Ένωση ε, είναι αρκετά σύντομες και ελπίζω να είναι και περιεκτικές. Για τεχνικούς λόγους λοιπόν είπαμε ότι οι προτάσεις θα είναι σύντομες. Ε, για ουσιαστικούς όμως λόγους έχω υποβάλει στα μέλη της Επιτροπής μία ε, πιο αναλυτική πρόταση για το τι θα έπρεπε να είναι οι εισηγήσει μας για την Ευρωμεσογειακή Ένωση στα πλαίσια της Ήτρε. Αυτό το οποίο το πρώτο που έχουμε ε, μπροστά μας, οι κωδικοποιημένες ε, προτάσεις, έχουμε την εισαγωγή η οποία κάνει αναφορά στις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ομπρέλα των οποίων μπορούν να αναλυφθούν οι διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις. Το θεωρώ σημαντικό λοιπόν να έχουμε ε, τις πολιτικές, πρωτοβουλίες όλα συγκεκριμένα που μπορούμε να αναφερθούμε για να μπορούμε να αναπτύξουμε δράσεις. Στην εισαγωγή προχωρούμε στην, στις υποδομές και στον εφοδιασμό όσον αφορά την ενέργεια, πάρα πολύ δικοποιημένα, όπου παραθέτω την αναγκαιότητα της ε, συντήρησης και ε, επέκτασης των δικτύων ενέργειας τόσο στο ε, αέριο, στο φυσικό αέριο όσο και στο πετρέλαιο κτλ. Ε, επισημαίνω την ε, μεγάλη σημασία και την ύπαρξη της ε, ηλιακής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και καταλήγουμε στο σημείο 4 με την ε, επίκληση για την θεσμοθέτηση μιας, ε, ενός κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τις επιχειρηματικές ε, δράσεις ε, στην περιοχή αυτή. Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η οικονομική συνεργασία είναι το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο θα μπορούσε ρεαλιστικά να οδηγήσει στην διαμόρφωση μιας ευρωμεσογειακής ε, ε, ενιαίας αγοράς ε, αγοράς υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. οι προτάσεις λοιπόν της Ήτρε θεωρώ ότι θα είναι καθοριστικές περισσότερο ίσως και από τις πολιτικές προτάσεις για το μέλλον της ευρωμεσογειακής συνεργασίας για το λόγο αυτό κύριε Πρόεδρε έχω συντάξει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες συνημένα σας έχουν διανεμηθεί και όπως είπαμε κάποιες από αυτές θα προωθηθούν ως ε, τροπολογίες στο τελικό κείμενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στην εισήγηση τη βασική που βλέπετε, αλλά υπάρχουν στο συνημένο κείμενο. Αυτές οι παράγραφοι του συνημένου κειμένου, κάποιες από αυτές είναι καθοριστικές για την ευρωμεσογειακή συνεργασία. Πολύ καθοριστικό θεωρώ το θέμα του LNG μια περαιτέρω διευκρίνηση με συγκεκριμένες προτάσεις για την ηλιακή ενέργεια, καθώς επίσης συγκεκριμένες προτάσεις και για την συνεργασία του επιχειρηματικού κόσμου και του εμπορικού κόσμου. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, τονίζω το εξής. Η εισήγηση είναι σύντομη, η βασική, αλλά θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να επικεντρωθούμε και στο συνημένο κείμενο που έχει πολύ ουσιαστικές προτάσεις πρώτον και δεύτερον θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να έχουν κατά νου ότι ορισμένες από τις παραγράφους του συνημένου κειμένου θα τις υποβάλω ως ε, τροπολογίες ε, στο τελικό κείμενο και θα ήθελα τη στήριξή τους γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και για το ότι μιλήσατε με τόσο συνεκτικό τρόπο και ε, συντάξατε και την έκθεσή σας επίσης με ευσύνοπτο τρόπο, γιατί ξέρετε έχουμε κάποιο πρόβλημα χρόνου και μας βοηθάει αυτή η ακρίβειά σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους ε, που βρίσκονται στην αίθουσα κατά πόσον θέλουν να λάβουν το λόγο, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, να κάνουν κάποια παρατήρηση. Η κυρία Κόμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, σαν σκιώδη συγγήτρια για το ΕΛΚ, όπως το είπε και η συγγήτρια, θα πρέπει να προωθήσουμε ιδιαίτερα συγκεκριμένε προτάσεις γιατί η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει μια κατάσταση με δυσκολίες οικονομικές. Είναι σημαντικό λοιπόν μια παρότριση με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής καταστάσεως και με διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων γιατί με τις πρώτες ύλε που είναι ένας πλούτος στην περιοχή της Μεσογείου ενδεχόμενα και να συντονίσουμε καλύτερα τα ε, οικονομικά όργανα όπως ε, την Τρέπεζα, την ευρωπαϊκή με ένα ταμείο κονδύλια ειδικά για τη Μεσόγειο και σε πλαίσια μια συνεργασία ανάμεσα σε περιφερειακά όργανα και τοπικά όργανα στην περιοχή της Μεσογείου. Συμφωνώ απόλυτα με τις υποδομές και την ανάπτυξή τους που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια. Σημαντικό όμως επίσης και μια υποδομή τηλεματική και πληροφοριακή για καλύτερη συνοχή με μια ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και της αγοράς γενικότερα στην ευρωμεσογειακή περιοχή. Όλα αυτά μπορούμε να τα διευκολύνουμε μέσω μεθόδων εμπορικών. Θα τα ευκρίσουμε αυτά με διάφορες τροπολογίες. Επαναλαμβάνω για τη διευκόλυνση αυτών των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Δεν βλέπω κανεί άλλο να ζητάει το λόγο. προ το πράγμα του... Α, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, δεν σα είδα. Ο συνάδελφο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τη στηρίξουμε γιατί αυτός ο χώρος της Μεσογείου έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό για τη συνεργασία των πολιτισμών ε, και οι αφρικανικές ε, εταιρείε μέσα από τις εμπορικές ανταλλαγές μπορούν να απτύξουν και άλλου είδους επαφές. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι το ευρωπαϊκό κομμάτι της ε, Μεσογείου αυτό το κομμάτι βεβαίως και παρουσιάζει διαφορετικά στάδια ανάπτυξης όσον αφορά την υποδομή των χωρών και την τεχνολογία. Ας πούμε, Έχουμε την Ιταλία, έχουμε τη Γαλλία, αλλά έχουμε και χώρες στα Βαλκάνια που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες. Ως εκ τούτου, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το σύνολο αυτών των χωρών, για αυτό το χώρο, θα μπορούσε να βοηθήσει κατά πολύ την περαιτέρω ανάπτυξη της ε, περιοχής. Πρόκειται για μια καλοσχεδιασμένη, σχεδιασμένη, συνετή πρωτοβουλία ε, και πρέπει λοιπόν τα βήματα που προτείνονται να στηριχθούν και μετά από τα λόγια να ακολουθήσουν και τα έργα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν νομίζω πια ότι θέλει κανείς άλλο το λόγο και νομίζω αυτό ισχύει πλέον. Κυρία Τζαβέλα, εσείς θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι. Να σας δώσω το λόγο. Πολύ ωραία. Ε, θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω θερμά και να επισημάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι 23η Μαρτίου 12 η ώρα είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών. Και να επισημάνω επίσης ότι όπως ε, συμφανίσαμε όλες οι τροπολογίες θα κατατεθούν στα αγγλικά. Και η... Ε, ο λόγος είναι πολύ απλός. Ε, υπάρχει μια ε, καταληκτική ημερομηνία που ορίστηκε από την ε, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή και για να μπορέσουμε να προλάβουμε πρέπει να τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση, δηλαδή η τροπολογία στα αγγλικά μέχρι τις 23 Μαρτίου και μετά ε, μπορούμε να ε, συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνει λοιπόν και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και πάμε στο επόμενο που είναι το υπαριθμό 6. Πρόκειται για την ε, συζήτηση με τον νέο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, είναι ο κύριος Φίλιπ Λόου τον οποίο και αναμένουμε από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, λέει ο Πρόεδρος. Ähm, Κύριε Λόου, ε, σας καλωσορίζω θερμά και χαίρομαι πάρα πολύ ε, που λίγο μετά την ανάληψη των ε, καθηκόντων σας ε, είπατε ότι θα έρθετε να μας επισκεφθείτε. Χαιρετίζω και τη συνεργατιδά σας και χαιρόμαστε που μπορούμε να κουβεντιάσουμε σήμερα. Βεβαίως... Θέλω να πω το εξής. Λυπάμαι πάρα πολύ που ε, μειώθηκε ο αριθμό των συναδέλφων που παρήσανται στην αίθουσα. Το λέω καταρχήν ε, για να γραφτεί στα πρακτικά. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι και φιλικό απέναντί σα. Γιατί να έρχεται τώρα εδώ ο Γενικό Διευθυντή για ένα θέμα που μα καίει και πολύ λίγοι παρόντε. Ε, Επίση, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι εσείς ήρθατε για να μας μιλήσετε. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι που είναι παρόντες θα εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα που τους προσφέρετε να κάνουν πολλές ερωτήσεις. Ε, εσείς βέβαια έχετε το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να ξεκινήσετε πρώτος και ε, μετά θα ακολουθούσουν οι άλλοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινούμε με αυτή τη συνάντηση μια νέα εταιρική σχέση, μια σχέση συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπή σα λοιπόν και τη νέα Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια. Πολλά έχουν γίνει ήδη στο παρελθόν, στον προηγούμενο σχηματισμό τη Γενική Διεύθυνση για να ενισχύσουμε την πολιτική ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με του συναδέλφου μου από την προηγούμενη Γενική Διεύθυνση, την Γενική Διεύθυνση Τρέν και την, το ε, πρώην Επίτροπο Πιμπάλξ. Ε, με το προσωπικό του και με τη σειρά μου τώρα εγώ θα σας προσφέρουμε ό,τι βοήθεια χρειάζεται ώστε μαζί να σχεδιάσουμε ένα τόσο σοβαρό χαρτοφυλάκιο και για όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασφαλή, διαρκή, καθαρή και από άποψη πόρων αποδοτική ενέργεια σε τιμή προσιτή και ανταγωνιστική. Προσπάθησα σε μια πρόταση να συνοψίσω τους στόχους της πολιτικής μας και ελπίζω ότι κανείς δεν θα εκπλαγεί εάν αυτή την πρόταση την επαναλάβω πολλές φορές τα επόμενα 3-4 χρόνια. Θα ακούσατε τον ε, Επίτροπο Έρτινγκ στι ε, ακρόαση, ο οποίος έκανε κάποιες προτάσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις που προβλέπουμε στην πολιτική μας. Εδώ θα ήθελα εγώ να επισκοπήσω τις πρώτες τι προκαταρκτικέ μα ιδέε για το πρόγραμμα εργασία για το 2010 και τα ερχόμενα χρόνια. Και επίση να πω και λίγα λόγια για το πώ ε, έχουμε οργανωθεί σε επίπεδο Γενική Διεύθυνση Ενέργεια προ στιγμή. Πρόεδρε, ήδη είχαμε πολλέ διμερεί επαφέ με μέλη τη Επιτροπή σα. Ελπίζουμε ότι θα τι ε, εξακολουθήσουμε. Όμω, εξίσου σημαντικό είναι να ερχόμαστε να μιλάμε και στο σύνολο των μελών τη Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εξισορρόπηση διαφορετικών απόψεων από αυτό χρειάζεται. Πράγματι, η νέα Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά της με μια δήλωση για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί ή πώς θα θέλαμε να έχει γίνει πλέον η Ευρώπη ως το 2020. Θα επανέλθουμε στο θέμα της ε, εξυπνής οικολογικής και από άποψη πόρων ευθυούς ε, κοινωνίας και οικονομίας, αλλά για να πετύχει αυτή η στρατηγική πρέπει να κάνουμε πολλά στο επίπεδο της ενέργειας. Ετοιμάζουμε τώρα ένα πρόγραμμα δράσης για την ενέργεια. Νομίζω ο κ. θα χρησιμοποιούσε τον όρο στρατηγική, γιατί πρόκειται πραγματικά για μια νέα στρατηγική, δεν είναι απλώς ένας κατάλογος μέτρων, και εκεί θα περιλαμβάνονται χειροπιαστά συγκεκριμένα μέτρα που σκοπεύουμε να λάβουμε για να επιδιώξουμε τους στόχους που ορίζονται τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Συγκεκριμένα, θέλουμε μια εύρυθμη και ανταγωνιστική ενιαία αγορά ενέργειας, αλλά και εν ώψη της ερχόμενης δεκαετίας θέλουμε να πετύχουμε και τους ε, στόχους 20-20-20 στο πακέτο των κλιματικών αλλαγών ή των μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύουμε ότι αυτή συνολική, αυτό το συνολικό πρόγραμμα δράσης για την ενέργεια θα εγκριθεί πλήρως το 2011. Ίσως ρωτήσετε γιατί δεν υποβάλαμε το πρόγραμμα αυτό ήδη φέτος. Πρώτον, πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις, ε, κατά κύριο λόγο μαζί σας, αλλά και με τους ευθύνοντες των κρατών μελών και όλους τους ενδιαφερομένους και γι' αυτό σκοπεύουμε τη διαδικασία να την εκκινήσουμε ετοιμάζοντας ένα, μια ενδιάμεση έκθεση, ντοκιμόντε τάπ όπως λέγεται, για το Συμβούλιο Ενέργειας τον Μάιο. Έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια ενδελεχή και προσεκτική μελέτη της στρατηγικής που περιέχει το πρόγραμμα προτού την, ε, πριν την έγκριση του μάλλον στις αρχές του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς η Επιτροπή σας θα διδραματίσει ζωτικό ρόλο στις σχετικές συζητήσει. Όπως και ο Επίτροπος νομίζω κατέστησε σαφέ κατά την ακρόασή του, δεν προτίθεται να ετοιμάσει ένα μακροσκελή κατάλογο με νέε νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ των προτεραιοτήτων μας στο να λειτουργήσει καλύτερα το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Άρα, όχι μόνο το τρίτο πακέτο, αλλά και το δεύτερο πακέτο μέτρων για την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλα αυτά. Να αναφέρω απλώς το ζήτημα της ανάπτυξης κωδίκων για την διασύνδεση των δικτύων μας. Θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση στην αγορά και για την προμήθεια στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, τους πολίτες με τους καλύτερους ενεργειακούς πόρους, αλλά και για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της προμήθειας. Της προσφοράς επίσης, συζητούμε ήδη την ε, ασφάλεια της προμήθειας σε φυσικό αέριο με σχετικό κανονισμό που μελετούμε επίσης πολύ εντατικά. Επιπλέον και για να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογικές λύσεις που είναι απαλλαγμένες από την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα εντάσσονται στις προτεραιότητες για την εξάλληψη του άνθρακα. Ε, μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων και μαζί με το πρόγραμμα δράση, ε, έχουμε συνεργαστεί στι υπηρεσίε τη Επιτροπή για να ετοιμάσουμε έναν οδικό χάρτη για την απαλλαγή των ενεργειακών μα πόρων από τον άνθρακα. Χρειάζεται βέβαια εντατική δουλειά για να φτάσουμε στου στόχου και σημαντικέ ενιστώσει αυτού του προγράμματο είναι κατά κύριο λόγο η απαλλαγή των μεταφορικών ε, μέσων και λύσεων από το διοξείδιο του άνθρακα. Να μια από τι πρώτε προτάσεις λοιπόν της Επιτροπής από την πλευρά της ενέργειας τώρα για τι υποδομέ και την ενίσχυσή τους. Το αναφέρατε Πρόεδρε και εσεί και οι συναδελφοί σας μόλι τώρα στα... στην όλη συζήτηση για την ε, Μεσόγειο, την περιοχή της Μεσογείου. Μας ενδιαφέρει και το δυναμικό και οι δυνατότητε για νέε λύσει στη Βόρεια Θάλασσα, την Βαλτική, τη Μεσόγειο αλλά και ανατολικά κυριως νοτοανατολικά, νότιο-ανατολικά σε, αυτήν την, σε αυτόν τον διάδρομο, την γεωγραφική ζώνη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αργότερα, μέσα στη χρονιά και παράλληλα με τις εργασίες μας για το πρόγραμμα δράσης, για την επόμενη πενταετία και δεκαετία, γνωρίζετε ότι θα υποβάλουμε και ένα πακέτο για τις ενεργειακές υποδομές. Εκεί θα εξετάζονται όλες οι επενδυτικές ανάγκες οι προτεραιότητε για τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου, η διαφοροποίηση τη προμήθεια και η κατάλληλη πρόσβαση για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Βεβαίω εδώ θα γνωρίζουν πολλά από τα μέλη τη Επιτροπή σα ότι είναι σημαντικό και το θέμα τη χρηματοδότηση. Όχι μόνο το επίπεδο τη χρηματοδότηση, ούτε η αναλογία απλώ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τα επιμέρου προγράμματα στη χρηματοδότηση. Γενικότερα η σημερινή οικονομική κατάσταση ε, μας ασκεί σοβαρές πιέσεις σε εμά και στις αγορές ώστε να φέρουν τα προτούμενα αποτελέσματα και προκειμένου να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Για προς το παρόν σε πολλές περιπτώσεις και περιοχές δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εμπορικά κίνητρα. Θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο να αναζητήσουμε την κατάλληλη συμβολή. Κατά τρίτον, αναφέρω το ζωτικό ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Υποσχεθήκαμε, εμείς και ο Επιτροπός μας βεβαίως, αναθεώρηση του ισχύοντος ε, προγράμματος δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ο σκοπός μας είναι να ε, υποβάλουμε όσο δυνατόν συντομότερα μετά από αυτό ένα νέο πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακριβώς ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, Ίσως είναι καλό να τα συνενώσουμε τα δύο αυτά ως ένα κοινό πακέτο, αντί να αποδυναμώσουμε την στατηγική σημασία των εγγράφων χωρίζοντάς τα σε δύο φάσεις. Πάντως, όπως έχουμε ήδη υποσχεθεί, ελπίζουμε ότι η αναθεώρηση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμεινο της χρονιάς και ότι οι προτάσεις για το νέο πακέτο θα γίνουν ως το δυνατόν συντομότερα μετά, το αργότερο στις αρχές του 2011. Κατά τα άλλα, έχω υπογραμμίσει νομίζω την σημασία της υλοποίησης της υπάρχουσας νομοθεσίας. Θα ήθελα να θυμίσω και τη σημασία της περάτωσης της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης ως προς την ενέργεια. Σε μεγάλο βαθμό έχουμε ήδη αποδεσμεύσει κονδύλια για προγράμματα που είχαν ε, θεωρηθεί προγράμματα προτεραιότητας Τώρα όμως θα πρέπει να δούμε και τι είναι εφικτό για το μικρό περιθώριο των μη δαπανηθέντων κονδυλίων που μας απέμειναν. Αυτό θα είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον της όθησης που θέλουμε να δώσουμε σε πολλούς νέους τομείς, την αιωλική ενέργεια και άλλες μορφές ενέργειας που θέλουμε να προωθήσουμε. Όσοι παρακολουθήσατε τις εξελίξεις για το τρίτο πακέτο της εσωτερικής αγοράς, θα γνωρίζετε ότι έχουμε και μια θεσμική πρόσκληση, πρόκληση εδώ να αντιμετωπίσουμε. Να δημιουργήσουμε σύντομα ένα ρυθμιστικό οργανισμό, η οποία θα διαμεσολαβεί, θα διαμεσολαβεί και θα επιλύει τα ζητήματα εσωτερικών διαφορών για την αγορά φυσικού αερίου. Εκεί θα συνδυάσουμε τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των εθνικών φορέων και σκοπό έχουμε να διορίσουμε διευθυντή αυτού του οργανισμού γύρω στα μέσα Απριλίου. Όπως θα γνωρίζετε, ο οργανισμός αυτός θα λειτουργεί στη Λιουμπλιάνα. Και ελπίζουμε ότι με τα μέτρα που τώρα προβλέπονται θα μπορέσουμε να επανδρώσουμε τον οργανισμό με το απαραίτητο προσωπικό, περίπου 50 άτομα. Και με την αρμοδιότητα, μάλλον με την ευθύνη, ως το Μάρτιο του 2011 να λειτουργεί πλήρως και αποτελεσματικά ο οργανισμό αυτό. Επίσημη ημερομηνία θέση σε ισχύ του τρίτου πακέτου για την εσωτερική αγορά. Βεβαίω, θα συνεχίσουμε την προετοιμασία για πολλά από αυτά που θα αναλάβει ο οργανισμό αυτό ήδη νωρίτερα και σε συνδυασμό με του εθνικού φορεί. Πρόεδρε, δεν θέλω να επεκταθώ στην εσωτερική διοργάνωση της γενικής μας διεύθυνσης θα γνωρίζετε ότι, και θα καταλαβαίνετε ότι σε σχέση με τις πολιτικές αποφάσεις της Επιτροπής να διαχωρίσει σε δύο σκέλη την πρώην Γενική Διεύθυνση Τρέν, μεταφορές και ενέργεια δηλαδή, όλα αυτά έγιναν με μεγάλη ταχύτητα. Αναζητήσαμε την τέλεια οργάνωση και στι δύο πλευρέ βεβαίω, αλλά ο Ματία Χούταρ και εγώ μπορέσαμε με τη βοήθεια των συναδέλφων μα να φέρουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Δεν λέμε ότι ο διαχωρισμό τη Γενική Διεύθυνση σε δύο ήταν απόλυτα αρμονικό και τέλειο. Κάποιοι πάλι πίστευαν ότι θα πάνε στι μεταφορέ και κάποιοι στην ενέργεια και πολλέ φορέ συνέβη το αντίστροφο. Όμω, ήδη έχουν ληφθεί απαραίτητε αποφάσει. Πιστεύουμε ότι το προσωπικό μα είναι πολύ αφοσιωμένο και πιστό και αναγνωρίζει ότι ο διαχωρισμό τη Γενική Διεύθυνση Σκέλη μα δίνει την ευκαιρία να επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα στι ε, σημαντικέ πολιτικέ μα προτεραιότητε στου δύο τομεί. Υπάρχουν δύο σημαντικέ αλλαγέ που ενδεχομένω να έχετε δει στον χάρτη διοργάνωση, στο διάγραμμα διοργάνωση τη Γενική Διεύθυνση Ενεργεία σε σχέση με το πρώην σκέλο τη Γενική Διεύθυνση Τρέν. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα στρατηγικό διευθυντή, ο οποίο συνδυάζει το έργο του παρατηρητήριου για την ε, ενέργεια και τι ε, διεθνεί συνεισφορέ. Και υπάρχει και μια υπηρεσία στρατηγική η οποία συνδυάζει όλες τις τάσεις και τις συνιστώσεις της ε, πολιτικής για την ενέργεια. Ελπίζουμε λοιπόν εκεί να υπάρχει συνεργασία, διάλογος, όχι μόνο με άλλους πολιτικούς τομείς που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με εξωτερικούς φορείς συμπεριλαμβανόμενες της ε, Επιτροπής σας. Ελπίζω ότι αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε έναν πιο αρμονικό και αποτελεσματικό ορισμό της ενεργειακής πολιτικής, άλλωστε υπάρχει και η συνθήκη της Λισαβόνας που μας υποχρεώνει σε κάτι τέτοιο. Το άλλο στοιχείο στο οποίο θέλω να δώσω έμφαση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει με ιδιαίτερη σαφήνεια τα σημεία, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον γερμανικό όρο, για τον διαχωρισμό εσωτερικού και εξωτερικού έργου χάραξης πολιτικής. Σημαίνει αυτό ότι η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαχείριση από την ίδια τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, οπότε αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την υπηρεσία ενέργειας τη ΡΕΛΕΞ στην Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Βαλτεμέρα και η διαδοχός του κυρία Άστον δεν θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά. Όμως, πρόθεσή μας είναι να δώσουμε μια συνεκτική ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή πολιτική κοινό. Δεν γίνεται να έχουμε ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια χωρίς να συνδυάσουμε τον το εξωτερικό σκέλος με το εσωτερικό. Την εξασφάλιση της προμήθειας δηλαδή, αλλά και εσωτερικά ποια είναι το σωστό ενεργειακό μείγμα και η εξισορρόπηση των αναγκών μας στον τομέα της έρευνας. Και εκεί ξεκινήσαμε, η Επιτροπή δηλαδή ξεκίνησε με τη δική σας στήριξη, πολλές νέες πρωτοβουλίες. Στον τομέα αυτό θα πρέπει να δώσουμε και άλλη όθηση. Θα πρέπει του χρόνου να συζητήσουμε το πόσο κονδύλια θα διατεθούν για όλα αυτά πριν το τέλος της αναθεώρησης του προπολογισμού. Θεωρούμε ότι οι επενδύσει σε νέους τεχνολογικούς τομείς για την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής αποτελεσματικότητα, είναι απαραίτητη, ζωτικότατη, προκειμένου να λειτουργήσει και αυτός ο τομέας. Η Επιτροπή δεν αποφάσισε από τώρα να συνδυάσει όλα τα διευθυντήρια έρευνα για την ενέργεια εντό τη Κομισιόν σε ένα. Κάποια παρέμειναν στη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και κάποια άλλα στη δική μα. Παρόλα αυτά, ο κ. Έτιγκερ ξεκαθάρισε ότι θα είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό για τα κονδύλια της ενεργειακής έρευνας. Συνεργαζόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή με τι αρμόδιε υπηρεσίε, ώστε ο Επίτροπό μα να έχει την πολιτική καθοδήγηση και διακυβέρνηση των διαφόρων αυτών τμήματων των ερευνητικών μα δραστηριοτήτων. Τέλο, ε, μερικά λόγια σε περίπτωση που κάποιοι σκεφτούν ότι το αμέλησα, η πυρηνική ασφάλεια και οι διασφαλίσει που χρειαζόμαστε. Αυτή είναι μια διαρκή προτεραιότητα. Έχουμε κάποια από τα καλύτερα πρότυπα και σύνολα των διαγραφών στην Ευρώπη και ο κύριος Έτιγκερ συνάντησε συναδέλφους μας στο Λουξεμβούργο για να συναντήσει το μέλλον της πολιτικής αυτής και από την άποψη της ασφάλειας και των διασφαλίσεων. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα φέτος με ένα σχέδιο οδηγίας για, την, ε, για τα πυρηνικά απόβλητα για την επεξεργασία του. Και αυτό θα είναι μια σημαντική συνιστόσα τη ε, Ευρωπαϊκή συνεισφορά στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Δεν είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι για τα πυρηνικά, αλλά είμαστε υπεύθυνοι για τι προδιαγραφέ ε, για την πυρηνική ασφάλεια και τι πυρηνικέ ε, εξασφαλίσει που χρειάζονται. Ο κύριος Έτιγκερ λοιπόν πιστεύει ότι εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε γιατικό ρόλο παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω θερμά ήταν ε, μια σαφής, ε, ευκρινέστατη περιγραφή του ε, ποιος ακριβώς είναι ο επιμερισμός των εργασιών. Παρακαλώ, μπορείτε αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, Αναφέρετε πολύ σημαντικούς ε, στρατηγικούς ε, στόχους για τη γενική σας διεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Στη νέα ε, γενική διεύθυνση υπάρχουν κάποιοι, κάποιες διευθύνσεις, κάποιες υποδιευθύνσεις που διεκδικούν την αυτονομία. Αλλά είναι διαμφισβήτητο ότι στον 21ο αιώνα είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μια γενική διεύθυνση για την ενέργεια, τη στιγμή που η ενέργεια τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους πολίτες είναι ύψης της σημασίας. Έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Πρώτη ερώτηση ποιο είναι το καθήκον της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης ε, σε δύο σημαντικούς τομείς. Αύριο θα ψηφίσουμε για την ασφάλεια ως προς το φυσικό αέριο και επίσης και για τον φορέα σχετικά ε, ο οποίος εκπονεί ρυθμίσεις για θέματα ενέργειας. Εγώ δεν κατανοώ ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας σε αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, επιτήρηση, τον έλεγχο του εφοδιασμού ε, με ενέργεια. Εδώ στο θέμα αυτό η Γενική Διεύθυνση θα προβεί σε αναδρομικές αναλύσεις του τι ακριβώς συνέβη κατά το παρελθόν. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της ε, απελευθέρωσης ε, των ενεργειακών ε, οδεύσεων. Γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι στο μέλλον θα υπάρξει μείωση της τιμής ενέργειας. Στην Ουγγαρία όμως δημιουργήθηκε μονοπόλιο και αυτό προκάλεσε αύξηση της τιμής της ενέργειας. Εσείς στα προγράμματά σας προβλέπετε να εξετάσετε αναδρομικά το θέμα της ε, απελευθέρωσης. Ο κύριος Κάρινς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Η μία ερώτηση είναι η εξής. Εσείς ε, αναφερθήκατε στο νέο ε, δημοσιονομικό εργαλείο για την ε, βελτίωση της υποδομής. Και είπατε βέβαια ότι η χρηματοδότηση είναι ένα θέμα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και η δική μου ερώτηση είναι η εξή. Ε, η Γενική Διεύθυνση τι είδους προτεραιότητες ορίζει Υπάρχουν ε, προγράμματα υποδομής ε, τα οποία είναι εμπορικά βιώσιμα και άλλα που δεν είναι απαραίτητα βιώσιμα, είναι όμως ε, απαραίτητα για την ασφάλεια της ενέργειας, ένα στο μέσο που υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις στην Ευρώπη. Εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθούν χρήματα κυρίως ε, στις περιπτώσεις εκείνες όπου διστάζει ο ιδιωτικός τομέας για να καλύψει το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που είναι εμπορικά βιώσιμο και σε αυτό που είναι απαραίτητο στην Ευρώπη για την ασφάλεια. Ε, δεύτερη ερώτηση. Κοινή ενεργειακή πολιτική. Δεν νομίζω ότι αναφέρατε κάτι επ' αυτού, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ε, πώς ακριβώς βλέπετε αυτό το κίνημα προς το να υπάρξει μια κοινή πολιτική, κοινίως ε, κοινή προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς ε, εφοδιασμό από τρίτες χώρες. Η τιμή του φυσικού αερίου αρχίζει να μειώνεται και υποθέτω αυτό οφείλεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, στο ότι η Shell ανακάλυψε κάποιες ε, άλλες δυνατότητες ε, κοιτασμάτων αερίου και γι' αυτό μειώνεται η τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε απαραίτητα το ίδιο στην Ευρώπη. Τουλάχιστον στη δική μου τη χώρα, τη Λετωνία, η εταιρεία την οποία ελέγχει η Gazprom λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει ότι θα αυξηθούν οι τιμέ του φυσικού αερίου κατά 30%. Αυτό δεν συμβαδίζει με τη γενικότερη εξέλιξη. Ε, γι' αυτό λοιπόν όταν ε, εξετάζουμε τις περιπτώσεις ή η ευρωπαικη Ένωση ε, απευθύνεται σε μεμονωμένες χώρες με μία φωνή, με, με κοινή στάση, τότε έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Όταν απευθύνει σε κάθε κράτος μεμονωμένο, ε, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Λόε. Εξ ονόματος της ομάδας μου καλώς ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, τις εξηγήσει σας σε τόσο σημαντικά θέματα δικής σας αρμοδιότητας, όπως επίσης και για τη λειτουργία της γενικής σας διεύθυνσης και τη διάθεση που αναφέρατε για συνεργασία μαζί μας. Δύο ερωτήσεις για σας για το σχέδιο δράσης ενέργειας, ε, γιατί βλέπουμε ότι εμφανίζονται και εξαφανίζονται στα κείμενα της Επιτροπής αυτές οι ενέργειες. Τώρα σημειώσαμε ιδιαίτερα το δικό σας χρονοδιάγραμμα. Να σας πω ότι λυπούμεθα από την ομάδα μου, γιατί όλα αυτά έρχονται κάπως αργά. Τουλάχιστον όμως αυτή φορά να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που αναγγείλατε. Να σας πω ότι στο θέμα αυτό σας εμπιστευόμαστε δεύτερο συγκεκριμένο ερώτημα, κύριε Λόου. Αποφάσισε η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα για τα, την υποδομή του σχεδίου ανακαμψής οικονομικής και έχουμε τρία επίπεδα. Μαζί με τα 50 εκατομμύρια στον σχετικό άξονα είχαμε 116 εκατομμύρια ευρώ και κάτι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σχέδια ακριβώς για ανανόσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή επαρκεία. Εδώ λοιπόν αυτά τα 100 περίπου 16 εκατομμύρια πώς θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα κατανεμηθούν από πλευράς Επιτροπής, τι φρονεί σχετικά η Επιτροπή λοιπόν κυρία Νίπλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Ε, κύριε Γενική Διευθυντά, αφενός το βρίσκω σωστό και καλό το ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας θα είναι αρμόδια και για την εξωτερική πολιτική σε σχέση με την ενέργεια. Θυμάμαι ότι ήταν, όταν ήταν εδώ ο κύριος Οτιγκέρ στην Ακρόαση, όταν ήταν υποψήφιος, σε αυτή την ερώτηση απάντησε ότι ε, ο τομέας αυτός ε, της ενέργειας επεκτείνεται συνεχώς. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που η εξωτερική πολιτική για την ενέργεια είναι στις ε, δικές σας αρμοδιότητες. Ξέρω ότι θα πρόξουν πολλές και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Έχω μία ερώτηση για το πρόγραμμα Desertec και ερωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ακριβώς το εντάσσει στη γενικότερη εξωτερική της πολιτική για την ενέργεια, πώς το αξιολογεί το πρόγραμμα, τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει. Δεύτερη ερώτηση αφορά στην απελευθέρωση των εσωτερικών αγορών ενέργειας. Τον τελευταίο καιρό έγιναν πάρα πολλά πράγματα και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, που γνωρίζετε πολύ καλά, ε, προσπάθησε να απελευθερώσει την αγορά και μέσα από το πακέτο της κοινή αγοράς ενέργειας εμείς συμβάλαμε σε όλο αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσείς ε, πώς ακριβώς ε, παρακολουθείτε την ε, εφαρμογή των κανονισμών. Υπάρχουν κάποιες ενδιάμεσες εκθέσεις και αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι το εξής. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία κράτη έχουν την, ε, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στα χέρια τους, σε μονοπόλια. Δεν θέλω τώρα να το σχολιάσω αυτό, αλλά εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι κατά πόσον, ειδικά στις χώρες εκείνες όπου το κράτος, με νομικές βέβαια διατάξεις, ε, έχει, όπως σας είπα, μονοπωλιακές δομές, κατά πόσον η Κομισιόν προτίθεται κάτι να κάνει γι' αυτό ή θα το αφήσει ως έχει. Δεν ξέρω τώρα γι' αυτό που θα ρωτήσω αν είσαστε ο σωστό συνομιλητή, αλλά αναφέρομαι στι ε, συζητήσει ε, στην Κοπενχάγη για το κλίμα. Ποια είναι η στρατηγική της ε, Κομισιόν. Θα προχωρήσει στι επόμενε διαπραγματεύσει με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια κατεύθυνση που έχει χαράξει ή θα καταβληθούν προσπάθειες ή περαιτέρω εξελίξει να προσαρμοστούν λιγάκι. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίω είναι τα πιστοποιητικά εκπομπών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως οι Αμερικανοί είπαν ότι δεν προτίθενται να εισάγουν ένα παρεμφερέ σύστημα, τουλάχιστον εν ευθέτω χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον ή μήπως ε, θα πρέπει λόγω των ε, διεθνών εξελίξεων να αναθεωρήσουμε λιγάκι και εμείς τη δική μας θέση και να την προσαρμόσουμε. Ο συνάδελφος κύριος ε, Πάσκα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά μάλλον, ε, είναι γνωστό σε όλους μας ε, ότι πρέπει να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν εκατομμύρια νοικοκυριών που χρησιμοποιούν συσκευές ε, παλιών προδιαγραφών των 220 βολτ. Υπάρχουν πολλές ε, ηλεκτρικές ε, συσκευές ε, στο νοικοκυριό που δεν χρειάζονται όμως αυτά τα 220 βολτ υπάρχουν μετασχηματιστές όπου μπορεί να μειωθεί η τάση μέχρι και τα 12 βολτ. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει ποια είναι τα προγράμματα της Κομισιόν για τα νοικοκυριά. Γιατί ε, θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω η χρήση της ενέργειας. Υπάρχουν έρευνες σε αυτό τον τομέα. Γίνονται αναλύσεις έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι νέες προδιαγραφές όπου όπως σας είπα για τις ε, περισσότερες ε, ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμεύσει χαμηλότερη τάση. Αυτό ε, θα ήταν και περισσότερο ασφαλές για τα παιδιά και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε και περισσότερη ενέργεια. Ο συνάδελφος κύριος Βίμπα. Κύριε Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά. Ακούστε, θα πρέπει από τη στιγμή που θέλουμε να ξεκινήσει με νέα δυναμικότητα οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα γίνει με κοινέ πολιτικές, ε, με νέα, αποτελέσματα. Να έχουμε κάτι παρόμοιο δυνατό με αυτά αποτελέσματα, κάτι το κοινό. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ την ενέργεια της δυνατότητές της σε κάθε μορφή. Μια διαπίστωση με εξέπληξε ιδιαίτερα. Πάνω σε αυτό να σας υποβάλω ένα ερώτημα. Την τρομερή καθυστέρηση, να μην πω φτώχεια, των συνδυασμών ενεργειακά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύνδεσης μπορώ να πούμε, γιατί νέες ε, τεχνολογίες εολικές ε, στο βορρά, φωτοβολταϊκά στο νότο, από τη στιγμή που αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί και να πέρασει σε αυτούς τους τομείς. Ε, αυτό ήθελα να ξέρω. Περισσότερα πράγματα, οι δικές σας οι προθέσεις, ποιες είναι για να ξεπεράσετε την καθυστέρηση αυτή στην διασύνδεση που παρατηρείτε. Πολλά έχουν να κάνουν με αρμοδιότητες της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά επίσης ε, αυτό έχει να κάνει και με τη δική μας την Επιτροπή και τις δικές μας ανησυχίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και την απόδοση της ενέργειας. Με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών ε, πώς θα συνεργαστείτε και βλέπω ότι στην υποδομή, κυρίως στην σιδηροδρομική, και για τα έξοδα αυτά βλέπουμε συνεχώς να προστίθεται καθυστέρηση ενώ υπάρχουν πηγές από τις οποίες θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε ενεργεία. Συνδυασμό λοιπόν και συνεργασία ανάμεσα στη δική σας δυνική Διεύθυνση και στις μεταφορές ώστε να αλλάξει κάπως η ροή των πραγμάτων σε αυτά. Σιμάνσκι. Ναι, όσα είπατε. Πολλά υπόσχονται με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, τη Νέα και τα σχέδια υπόσχονται πολλά για την εξωτερική πολιτική αυτής της ε, πτυχή αυτής της ενεργειακής πολιτικής. Εδώ μιλάμε για διπλωματία, για εξωτερική πολιτική, πολλά και διάφορα που ανακατεύονται, μπερδεύονται και τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον θα είναι κάτι το ιδιαίτερα γοητευτικό ενδιαφέρον. Τι γίνεται με την ασφάλεια από τα ραδιενεργά απόβλητα και τι γίνεται με τον Έτρικερ, τον επίτροπο που θα επισκεφθεί την Πολωνία, η πρώτη επίσκεψή του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επίσκεψη αυτή θα ασχοληθεί με την Πένιγκιν και Γκάσπροπ και τις αντιφατικές ακριβώς λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτών των δύο. Εγκ, κύριε Εγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα, αλλά είχα δύο ψηφοφορίες σε δύο διαφορετικές επιτροπές προηγουμένως. Εκ μέρους της ομάδας Άλντε, ήθελα να σα καθορίσω θερμά. Βεβαίω, θα είσαστε ένα από τα πιο πλέον σημαντικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη, σε ό,τι θα αφορά βεβαίω την ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώ και του στόχου του 2020. Το να πιστέψουμε στην δυνατότητα αποταμίευσης και εξοικονόμησης ενέργεια, ενέργειας είναι σημαντικό και έχετε ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια σας και τους κλιματικούς στόχους και την στρατηγική για το 2020 εξοικονομήσει στην ενέργεια. Υπάρχει σαφής στόχος. Όταν λοιπόν λέτε ότι θα έχουμε το πρόγραμμα δράσης επιτέλους για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ελπίζω ότι θα προβλέψετε υποχρεωτικούς δεσμευτικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν βλέπουμε τι δυνατότητες υπάρχουν γι' αυτό. Μέχρι 200 δις ευρώ ετησίως θα μπορούσαμε να εξοικονομούμε και να δημιουργήσουμε και ένα μεγάλο ρυθμό θέσεων εργασία. Είναι λοιπόν ε, κορυφαία σημασία στο θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν να μας δώσετε μια ημερομηνία και τις απόψεις σας για τους στόχους. you. I also want to welcome you in the... Ο κ. Γόντε, ε, ήθελα να σας ε, καλωσορίσω στην Επιτροπή μας και όπως μόλις είπε και η κυρία Εκ, Νομίζω ότι όλοι ανυπομονούμε να δούμε το πρόγραμμα δράση για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αναθεώρησή του. Σημειώνουμε ότι η Επιτροπή σκόπευε ήδη από το περασμένο φθινόπωρο να δημοσιεύσει κάτι τέτοιο. Έχω τρει ερωτήσει. Η μία είναι ποια η γνώμη σα για το να γίνει υποχρεωτικό ο στόχο εξοικονόμηση ενέργεια κατά 20%. Δύο, Πώ η Επιτροπή θα συμβάλλει στο στόχο διασφάλιση ότι τα μη δαπανηθέντα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ανάκαμψη, την οικονομική ανάκαμψη, θα δαπανηθούν για προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τέλος, υπήρξαν κάποιες κινήσεις κερδοσκοπίας ή μάλλον κάποιες ε, υποθέσεις για το πώς θα ε, συνεργαστεί η Γενική σας Διεύθυνση με τη Γενική Διεύθυνση στην Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τις κλιματικές αλλαγές. Έχετε ίσως κάποιο αγώνα, κάποιο κοινό πρόγραμμα μάλλον συνεργασίας με την υπεύθυνη Γενική Διεύθυνση ή υπάρχει κόντρα μεταξύ σας, κόντρα εξουσίας για το ποιος θα αναλάβει τις αρμοδιότητες. Ευχαριστούμε ο κύριος Ζανό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον Γενικό Διευθυντή. Όπως είπε ο κύριος Σάκ, το προς αυτήν την κατεύθυνση και εγώ για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παντού όλοι συμφωνούν. Είναι σημαντικό για την προμήθεια, για την απασχόληση, για την οικονομία, για το κλίμα. Όλοι συμφωνούν. Και μας είπαν για το πρόγραμμα του 2009. Το έγινε 2010. Άντε το πήγαμε τώρα στις 2011. Τι κάναμε και μας λένε ότι θα έχουμε σούπερ σχέδιο για την ενέργεια, για την υποδομή επίσης. Ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, ειδικά προγράμματα, ειδικές δαπάνες, κονδύλια. Πεστε μου εσείς ε, έτσι πώς ε, ε, τι λέτε για αυτή την προσφορά χωρίς να σκεφτείτε και τη ζήτηση. Έχουν τρομερά ελλείμματα οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Τι γίνεται, πώς θα προχωρήσετε πριν να ξέρετε πόσο θα καταναλώσει κάνει. Σας ευχαριστώ που μας διαβεβαιώνετε ότι δεν θα, υπάρχουμε, δεν θα υπάρχει σχέδιο πρόγραμμα για την ενέργεια εάν δεν υπάρξει πρώτα για την ε, αποτελεσματικότητα μια βεβαίωση για το ε, ε, οικολογικό design είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε να κάνουμε με τους καυστήρες της, τη θέρμανση το 25% στην Ευρώπη θα είχαμε 44 δισεκατομμύρια ευρώ αν είμαστε φιλοδεξοί και 220 εκατομμύρια τόνοι μέχρι το 2020 κομπής δεξιού του άνθρακος είναι τρομερή ποσότητα αυτή. Τι γίνεται και ακούμε από την Γενική Διεύθυνση πολλές συχνά κάθε εβδομάδα να μας λένε ότι εντάξει απόδοση, αποθετικότητα ενεργειακή χαμηλότερη. Τι γίνεται, θα θέσετε ένα τέλος σε αυτά, τα πράγματα, σε αυτή τη μείωση φιλοδοξιών για να έχουμε αντίθετα ισχυρέ φιλοδοξίε ότι θα έχουμε και θα πραγματοποιήσουμε μεγάλες εξοικονομήσεις. Μαλονέσκο. Thank you, Chair. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Ήθελα να θέσω μία ερώτηση. Ποια η θέση του Ναμπούκο στην στρατηγική τη στρατηγική που προβλέπεται για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Και ποια η άποψή σας για τον αγωγό Ναμπούκο σε σχέση με το South Stream. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Είδατε πάρα πολλές και διαφορετικές ερωτήσεις σε διαφορετικού περιεχομένου ε, και προσπαθήστε τουλάχιστον να απαντήσετε. Ξεκινήσω εγώ. Τέθηκε μια σειρά από ερωτήσεις, ιδίω για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα πρέπει να σας πω ξεκάθαρα ότι έγινα πριν από 18 ημέρε, όχι μήνε, με συγχωρείτε, ημέρε, Γενικό Διευθυντή, φαίνεται σαν να ήταν 18 μήνε βέβαια, έτσι το αισθάνομαι. Αλλά η ημερομηνία που θα σα δώσω, μόλι την έχουμε ορίσει, θα είναι ο στόχο μα έτσι κι αλλιώ. Ξέρω ότι ο κύριο Έτιγκερ συμφωνεί μαζί μου. Στην περιοχή του ανταγωνισμού όμως, που έχω ήδη κάποια εμπειρία, μόλις δίνω ένα ραντεβού μια ημερομηνία, ισχύει πάντοτε. Και δεν το λέω αυτό μόνο από την πλευρά της Επιτροπής, αλλά για την συνολική πολιτική της, ευρωπαϊκής, της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι μια προσωπική δέσμευση αυτή. Πρέπει όμως να σας πω τώρα ποιο είναι το ρεαλιστικό μας χρονοδιάγραμμα και τι δεν είναι εφικτό. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα κάτι παραπάνω. Πρέπει να ζητήσω την υπομονή σας. Όμως, εφ' εξής, όπως σας ξαναείπα και εγώ και ο κ. Έτιγκερ ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει απλώς να επεξεργαστούμε, να το αποφασίσουμε και να σιγουρευτούμε ότι έχουμε τις σωστές προσδοκίες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όσα είπε ο κ. Ζαντό για την απελευθέρωση και όσα έχουν γίνει ως τώρα και αν ήταν επιτυχημένα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχουμε σοβαρή απελευθέρωση τη αγορά ενέργεια και τη αγορά φυσικού αερίου ακόμη. Ιδίω στι περιοχέ που αναφέρατε. Κυρίω βασιστήκαμε στη μελέτη που έκανε πριν από δύο χρόνια η Επιτροπή. Υπάρχουν εθνικέ αγορέ όπου δεσπόζουν πολύ σοβαροί, σημαντικοί φορεί και είναι δύσκολο να προσφερθεί περισσότερη επιλογή στους καταναλωτέ. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχολούν στην υλοποίηση του τρίτου πακέτου για την ενιαία αγορά είναι να ανοίξουμε τις, να πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητες των ε, πολιτών για την προμήθεια προϊόντων ε, σε περιοχές και περιφέρειες όπως η δική σας. Πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές για το ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές των προϊόντων σε αυτή την περίπτωση. Σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να έχει προϋπάρξει μια μακράς διάρκειας σύμβαση με το συγκεκριμένο παρέχοντα, προμηθευτή και για 30 χρόνια κάποιες φορές και οι συνθήκες αυτές είναι τόσο αποκλειστικές τόσο ιδιαίτερες, που θα είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε σε όλους ότι η άμεση επίπτωση της, του ανοίγματο των αγορών θα είναι επίπτωση των τιμών. Εάν δει βέβαια κανείς τη ζήτηση για την προσφορά γενικότερα στον κόσμο μας, δεν μπορούμε να πιστεύουμε ρεαλιστικά ότι θα επιτύχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε με τις τηλεπικοινωνίες ή τις αεροπορικές μεταφορές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αγορά που να είναι ανταγωνιστική, να προσφέρει ενέργεια ανταγωνιστικά με τιμές προσιτές, αλλά έχοντας κατά νου και τους στόχους για το διοξείδιο του άνθρακα. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι προϋποθέσεις υπάρχουν, ώστε οι επιχειρήσεις και οι κοινοί πολίτες, οι απλοί άνθρωποι να έχουν ε, ό,τι καλύτερο είναι δυνατό προϊόν. Δεν μπορώ όμω να αποκλείσω τι εξαιρετικέ αυτέ συνθήκε, όπου οι πρώτε επιπτώσει ε, για τι τιμέ, οι βραχυπρόθεσμε, θα είναι διαφορετικέ. Όμω αυτό που μα απασχολεί θα συμβεί μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, α πούμε ότι σε μια χώρα υπάρχει ένα ε, προμηθευτή για όλο το αέριο. Εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε καθόλου για απελευθέρωση. Δεν έχει υπάρξει απελευθέρωση. Εκεί πρέπει να επιβάλλουμε την απελευθέρωση τη αγορά. Να ποια θα είναι τα ζητήματα που θα απασχολήσουν το δεύτερο και τρίτο πακέτο. Ποιο ο ρόλο τη Γενική Διεθνή Ενέργεια εδώ. Η Επιτροπή όπω ε, την οδήγησαν οι προκάτοχοί μου στην πολιτική τη, έχει προτείνει τέτοια, τέτοια μέτρα για την απελευθέρωση τη αγορά αερίου. Ήδη η ομάδα συνεργατών μου συζητά τέτοια ζητήματα. Ποιο θα είναι λοιπόν ο σκοπό ενός ευρωπαϊκού κανονισμού για την παροχή φυσικού αερίου. Θα είναι να δούμε ποιες ε, καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, να πυροδοτήσουν την ελληνική ας πούμε, ώστε να υπάρξει προμήθεια φυσικού αερίου σε γείτονε χώρε. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε που μπορεί να προκύψουν καταστάσεις επίγουσες. Λόγω χάρη ένα πρόβλημα στις υποδομές μιας συγκεκριμένης χώρας κατά πόσον θα μπορούσαν αυτομάτως να βοηθήσουν οι γείτονες τη συγκεκριμένη περιοχή μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου κανονισμού. Βεβαίως πολλά θα εξαρτηθούν σε καθημερινή βάση από τη δράση και των ρυθμιστών και των εταιριών. Όμως μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο πραγματικά προσπαθεί να θεσπίσει βασικού κανόνε για το πώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπεριφέρονται και πώ κάθε κράτο-μέλο θα αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Η αλληλεγγύη θα είναι ένα καθοριστικό κριτήριο στο νέο και είναι στο καθοριστικό στοιχείο στο νέο άρθρο περί ενέργειας στην νέα συνθήκη. Το πώς λειτουργεί ως τώρα η αγορά και αν το έχουμε μελετήσει αυτό. Βεβαίως, βεβαίως ε, θα δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν, όπου δεν έχουν εφαρμοστεί λόγω χάρη σωστά οι κανόνες του δεύτερου πακέτου. Μας ενδιαφέρει να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη υλοποιούν τους κανόνες, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο για τη σταθερή προσφορά, ανταγωνιστικές τιμές επίσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, όπως είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των ρυθμιστών για το πόσο αέριο και πόσο ε, ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να περνάει από τη μια χώρα στην άλλη. Δεν είναι το ίδιο με τον τομέα των συντηροδρομικών μεταφορών. Εκεί είδαμε κάποιοι οδηγοί να φεύγουν από το τρένο και να κατεβαίνουν από την απομηχανή για να πάρει τα ενία κάποιο άλλο μηχανοδικό και να περάσει το τρένο τα σύνορα. Δεν είναι έτσι με την ενέργεια όμω, διότι οι εθνικοί ρυθμιστέ ω τώρα έχουν επικεντρωθεί στι εθνικέ ανάγκε των εθνικών δικτύων και φροντίζουν να ε, καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες σε εθνικό επίπεδο. Τα πλεονεκτήματα και σχέσεις συνεργασίας όμως ε, όλοι πρέπει να τα δουν χρησιμοποιώντας τέτοια συστήματα διασύνδεσης. Γιατί όμως δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες διασύνδεσης ήδη. Για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί εταιρείε και ρυθμιστές ουδέποτε έλαβαν υπόψη τα υπερεθνικά ωφέλη που μπορεί να έχει το να ξεπεράσει κανείς το εθνικό του δίκτυο. Για λόγους λοιπόν ασφάλειας της παροχής και για λόγους ανταγωνιστικότητας πρέπει να εξασφαλίσουμε την διασύνδεση των δικτύων. Τώρα για το ζήτημα των υποδομών. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικές. Πρέπει πρώτα απ' όλα όμως κανείς να διατηθεί σε τι επίπεδο και υπό ποιες προϋποθέσεις οι υποδομές που χρειαζόμαστε μπορούν να δημιουργηθούν. Για να απαντήσω με τρόπο απλό στο βασικό σας ερώτημα, ποια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, να σας πω ότι θα ήταν ανόητο οι δημόσιες αρχές να παρέμβουν σε τομείς όπου υπάρχει σημαντικό κέρδος εμπορικό ε, για να εξασφαλίσουν τη διασύνδεση. Εμείς θέλουμε να δούμε πού η αγορά δεν καταφέρει να φέρει τα απατούμενα αποτελέσματα και εκεί να παρέμβουμε. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι κάποτε εταιρείε θα κάνουν τι απαραίτητε επενδύσει, εάν δεν το κάνουν με αρκετή ταχύτητα, προκειμένου τα ωφέλη να τα αποκομίσουν όλοι οι πολίτε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, εκεί θα παρέμβουμε. Άρα θα εντοπίσουμε πέρα από, την από τον παραδοσιακό ορισμό των ανεπαρκειών ή ελλείψεων της αγοράς, που συμβαίνουν πράγματα που μπορεί να είναι κοινωνικά επιθυμητά αλλά εμπορικά με βιώσιμα. Και το θέμα είναι και το χρονοδιάγραμμα. Τι θα πρέπει να επιταχύνουμε λόγω χάρη, να επισπεύσουμε για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην ενεργειακή παροχή. Δεν μπορώ να σας πω ήδη από τώρα ποια θα είναι τα τελικά μας συμπεράσματα βεβαίως για αυτό το θέμα. Πολλές φωνές ακούγονται σε όλη την Ευρώπη, πολλές απόψεις εντός του τραπεζικού τομέα, μεταξύ των δημοσίων αρχών, λένε ότι αναπόφευκτα θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο κεφάλαιο χρηματοπιστωτικό σε συγκεκριμένα προγράμματα από δημόσια κονδύλια, ώστε να ξεκινήσουν επενδυτικές ενέργειες και δραστηριότητες που μπορεί να μην δίνουν τεράστιο κέρδος, αλλά είναι και χαμηλού κινδύνου. Εάν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα δημοσίων επενδύσεων, μέχρι των ε, χρηματιστηριακών αξιών και ως ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αυτό θα γίνει. Τώρα, με το χρόνο και αφόσον οι τιμές εξισορροπηθούν και ανέβουν, ελπίζοντας ότι θα αναπτυχθεί και το πρόγραμμα για τον έλεγχο των εκπομπών του άνθρακα, οι αγορές εν τέλει θα μπορέσουν να αναλάβουν και να αποκαταστήσουν ε, το ρόλο αυτό. Γιατί μέχρι το 2015 θα έχει και εμπορικό νόημα να επενδύει κανεί αυτά. Όμως ε, τώρα με τα προβλήματα που έχουμε με το αέριο και με την οικονομική ύφεση υπάρχουν, υπάρχουν ανησυχίες για τα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Δεν μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν ήδη σήμερα. Το ερώτημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο πλαίσιο το πακέτο για τις υποδομές αν ήταν εδώ ο κύριο Έτεγκερ και όταν ήταν εδώ, ανέφερε την ανάγκη να γνωρίζουμε σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Είναι κάτι που πανευρωπαϊκά θα πρέπει να το πράξουμε. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να αναλάβουν ε, δράση, να δώσουν τα θεσμικά όργανα κονδύλια ή να υπάρξει δικτύωση μεταξύ τους των δημοσίων αρχών στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες και τους παρόχους τους. Ναι, ο αγωγός Ναμπούκο είναι είναι πρόγραμμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει θερμά. Γι' αυτό γιατί. Γιατί σε σύγκριση με όλα τα άλλα που συμβαίνουν στην νότια γεωγραφική, στα νότια σύνορά μας, στην νότια περιοχή, σχέδια για τα οποία καταρχήν είναι θετική η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ έχουμε περισσότερα πλεονεκτήματα. Διαφοροποίηση των πηγών, πηγές διαφορετικές, όχι μόνο από το Τουρκμενιστάν και το Αζερβαϊτζάν, αλλά και από το Ιράκ και διαφοροποίηση της προμήθειας. Ελπίζουμε ότι το αγωγός θα, θα καταφέρει να δίνει ε, προϊόντα αερίου, να παρέχει αέριο σε ένα δίκτυο χονδρικών πωλήσεων πλέον. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα όμως, στον ίδιο νότιο διάδρομο, το ITGI και άλλα, το White Stream για το οποίο ο κ. Σέτιγκερ σκοπεύει να διοργανώσει μια διάσκεψη αλλά και για τον αγωγό Ναμπούκο αργότερα μέσα στη χρονιά ώστε να συζητηθεί κατά πόσο τα προγράμματα αυτά μπορούν να επισπευστούν. Ωστόσο, η Επιτροπή ήδη έχει στηρίξει θερμά το πρόγραμμα Ναμπούκο. Θεωρεί ότι συνδυάζει πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα και είναι κάτι στο οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Για το South Stream τώρα. Εδώ έχουμε άλλη κατηγορία πρόγραμμα. Αλλά δεν μα απασχολεί και λιγότερο. Εκεί βέβαια ο στόχο δεν είναι να ανοίξουν τα δίκτυα ούτε να διαφοροποιηθεί η προμήθεια. Απλώ η ίδια η ποσότητα αερίου θα περνάει πλέον όχι από την Ουκρανία αλλά από τον Νότιο Διάδρομο. Δεν έχει λοιπόν τέτοια στατηγικά πλέον εκτήματα όπως το Αμπούκο. Για το πρόγραμμα δράσης τώρα και το χρονοδιάγραμμά μας. Κοιτάξτε, πρέπει να πω κάτι όπου ως ε, στέλεχος της Επιτροπής είναι περίγοντο λέει κανείς τους πολιτικούς της Επιτροπής σα είναι εύκολο να έχει κάνει καταληκτική ημερομηνία για ένα πρόγραμμα δράση. Αλλά είμαι ότι όταν είχε υιοθετηθεί ήδη το πρόγραμμα δράση της Επιτροπής ε, από το 2009, πριν τι εκλογέ του Ευρωκοινοβουλίου, πολλοί θα μα είχαν πει για περιπέντε. Αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να συζητηθεί με λεπτομέρειες με το Κοινοβούλιο πριν κυρωθεί Γι' αυτό λοιπόν, πρωτού εγκρίνουμε πρόγραμμα δράση που θα καλύπτει όλα όσα θέλουν να κάνουν ο κ. Σέτιγκερ και η Επιτροπή στο 2013, αλλά θέλει να θέσει και στόχου και για το 2020, δηλαδή θα θέσει τι βάσει. Θα σχεδιάσει ολόκληρο το σκηνικό και θα κινητοποιήσει σοβαρέ δραστηριότητε για του τομεί που μα απασχολούν, μέτρα εσωτερική αγορά, υποδομέ. Όλα αυτά απαιτούν μακρόπνοη δράση και φιλόδοξου στόχου και εντατική δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την περίοδο συζητήσεων. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαστήκαμε να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να εγκριθεί μετά από έξι μήνε. Αυτό είναι και ο λόγο λοιπόν που ακολουθήσαμε αυτή την πολιτική γραμμή. Και εγώ και ο κύριο Έτιγκερ. Πέραν αυτού, είμαι σίγουρο ότι θα έχετε να πείτε πολλά και να σχολιάσετε πολλά για όσα θα ετοιμάσουμε. Όμω, ε, το χρονοδιάγραμμα που έχω εγώ στα χέρια μου για να ετοιμάσω αυτό το πρόγραμμα δράση είναι σαφέ. Μια πρώτη μορφή του προγράμματος όμως. Αν σας έλεγα ότι θα ετοιμαστεί το Μάιο, σημαίνει ότι θα πρέπει να το έχω ήδη σχεδόν ολοκληρώσει σε τρεις εβδομάδες. Πάντως να είστε βέβαιοι, θα έχετε το χρόνο και να το δείτε και να αντιδράσετε. Και να επανέλθω τώρα στο Desert Tech. Και εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε στηρίξει καταρχήν και το οποίο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες. Όμως θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό θα πρέπει εδώ να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και κατά πόσον θα μπορέσει να διασυνδεθεί με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό σύστημα. Για την Κοπενχάγη και τι άλλαξε. Η αλλαγή τώρα είναι ότι η ενεργειακή πολιτική στο παρελθόν θεσπιζόταν και καθοριζόταν χωρίς διεθνή συμφωνία για τις προτεραιότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τώρα, στην Επιτροπή, αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται περισσότερη περικοπή των εκπομπών σε 30% και υπό την πρωτοβουλία της αρμόδιας επιτρόπου συμφωνήσαμε να δούμε και τι είναι αναγκαίο να γίνει για να επιτύχουμε το στόχο των 30%. Χωρί όμω να ληφθεί και επίσημη απόφαση, λόγω και των διεθνών εξελίξεων. Νομίζω όμω ότι και άλλοι επίτροποι, ιδίω ο κ. Έτιγκερ, θα έλεγαν και πιστεύω ότι και οι γνώστε για το κλίμα θα συμφωνούσαν ότι ο στόχο τη ενέργεια δεν απλώ να σωθεί στον κόσμο και δεν παράγουμε ενέργεια και ενέργεια πολιτικής, πολιτική μάλλον ενέργεια μόνο για σκοπούς φιλανθρωπικούς, αλλά και για τους εμπορικούς μας λόγους, για να δώσουμε ενέργεια στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, για να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν απλώς να διστάζουμε και να λέμε ότι χάσαμε το ρυθμό των εξελίξεων απλώς γιατί δεν πήγαν καλά τα πράγματα στην Βεβαίω και πρέπει να διαφοροποιήσουμε την προμήθεια ενέργεια στην Ευρώπη. Είναι λογικό αυτό. Πρέπει να βασιστούμε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Η Κίνα και η Ινδία το κάνουν αυτό. Εμεί τι θα λέμε, ότι επειδή ανησυχήσαμε για την Κοπενχάγη και στενοχωρηθήκαμε με τα αποτελέσματα, θα χάσουμε το ρυθμό μα. Ναι, σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρξει κάποια άμεση εμπορική κινητοποίηση, ούτε θα δοθούν κίνητρα εμπορικά αμέσω ώστε ως προς τις νέες τεχνολογίες και τις υποδομές όλα να προσφερθούν απλόχερα. Όμως, εμείς έτσι κι αλλιώς θεωρούμε ότι περνάμε από μια μεταβατική περίοδο. Ένα τέτοιο φαινόμενο και θα πρέπει να αντέξουμε σε αυτή την περίοδο που γνωρίζουμε ότι η συνεργασία μεταξύ των μεγαλύτερων συμμαχιών ε, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να δώσουν αποτελέσματα. Πάντω, όπω βλέπετε και για τη στρατηγική του 2020, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν μέσα ε, που να βασίζονται στην αγορά και για τα πιστοποιητικά που θα χρειαστούν και για τις δράσεις, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος μας δεν είναι απλώς να θυσιάσουμε τους πολίτες της Ευρώπης και τις εταιρείε της Ευρώπης για κάποιον άγνωστο σκοπό. Θέλουμε να επιδιώξουμε συγκεκριμένους στόχους, βεβαίως, αλλά βασική μας στρατηγική θα πρέπει να προσαρμοστεί για την ενεργειακή αποδοτικότητα και πάλι. Θα πρέπει να περάσουμε από την ε, αναθεώρηση της οδηγίας για τις υποδομές, για την ατικετοθεσία επίσης. Όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν στην περάτωση του πακέτου, του σχετικού πακέτου. Δεν μπορώ να σας δώσω μια οριστική απάντηση για το αν τα πάντα στο πακέτο ενεργειακή αποδοτικότητα θα μπορούσαν ε, να οριστούν σε βάση υποχρεωτική ή εθελούσια. Πιστεύω ότι σε πολλού τομεί και αυτή την απόφαση θα τη λάβει η Επιτροπή, το εάν θέλει να ορίσει υποχρεωτικού στόχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω λοιπόν ότι ένα πράγμα είναι σαφέ Ότι υπάρχουν μέτρα τυποποίηση και μέτρα αριθμιστικά, τα οποία πρέπει να αναλυθούν πάση θυσία, προκειμένου να ε, τονώσουμε την επιχειρηματική πρωτοβουλία στην ενεργειακή υποδοτικότητα. Η ευφυής μέτρηση, τα τεχνικά μέτρα, οι ειδικέ ε, τεχνικές προδιαγραφές χρειάζονται περαιτέρω διευθέτηση για να λειτουργήσουν. Αυτό θα είναι σαφώς μια συνιστόσα του πακέτου για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όμως είχε πει και ο κ. Έτιγκερ στην ακρόασή του αυτό θα πρέπει να βασιστεί σε μια εταιρική σχέση μεταξύ των όσων πράγματι είναι υπεύθυνοι των τοπικών, περιφερειακών και επιμέρους πρωτοβουλειών για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε κτίρια και νοικοκυριά. Δεν νομίζω κανείς να προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει τα υλικά στους πολίτες για να μονώσουν τις στέγες τους. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες αρχές. Πάντως, την επιλογή μεταξύ υποχρεωτικών ή εθελοντικών μέτρων την αφήνω ανοιχτή. Σίγουρα υπάρχουν τομείς, όπως ο τομέας των... του επίπεδου της προσφοράς ή των φωτοβολταϊκών. Ναι, εκεί χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση, για να είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα λειτουργήσουν έμπριθμα η δική μου η εντύπωση για τους ευφύς μετρητές λόγου χάρη είναι ότι ως τώρα αυτοί έχουν ωφελήσει τους, ε, τις εταιρείες ενέργειας, πώλησης, ε, προσφοράς ενέργειας δηλαδή και όχι τους καταναλωτές. Θα τα δούμε όμως αυτά. Θα δούμε κατά πόσον χρειάζεται μια επιστροφή στο δίκτυο. Αν απλώς υπάρχει όφελος όμως για τις επιχειρήσεις και κανένα κίνητρο για τους ανθρώπους να εξοικονομούν ή να στραφούν στις ανανεώσιμες πηγές, κάτι που θα ήταν για τους ίδιους επικερδές δηλαδή, τότε δεν θα έχουμε τα σωστά κίνητρα. Κάποιος επίσης είπε και ρώτησε εάν θα συνεργαστείτε με τους συνεργάτες σας, τους ε, συναδέλφους σας στην Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Το παράθυρο όμως στον ίδιο όροφο, στον 8ο όροφο δηλαδή, με την παλιά διεύθυνση Τη γενική διεύθυνση, με, την παλιά, μάλλον, με τα παλιά γραφεία τη Γενική διεύθυνση Τραν, ε, όπου τώρα βρίσκονται τα γραφεία τη Γενική διεύθυνση Μεταφορών. Εγώ μπορώ να χαιρετήσω τον απέναντι συνάδελφό μου κάθε μέρα, από το παράθυρό μου. Έχουμε κοινέ υπηρεσίε, παρόλο που προσλάβαμε και περισσότερο προσωπικό για να επαντρώσουμε τι δύο γενικέ διευθύνσει. Δεν θα σα εκπλήξει το γεγονό ότι εκτό από καλοί φίλοι και συνάδελφοι, είμαστε και αναγκασμένοι να συνεργαστούμε με τον Ματία Γκουτ. Το θέμα λοιπόν της απαλλαγής των μεταφορικών μέσων από τον άνθρακα είναι πάντοτε περίπλοκο, είναι ευαίσθητο, γιατί έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Για την ηλεκτρική ενέργεια τον απαλλαγούμε από τον άνθρακα δεν είναι απλό. Ούτως ή άλλως η ενέργεια και αποδοτικότητα είναι ένας τομέας δύσκολος. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συμπεριφορά των πολιτών ατομικά, αλλά για τα ηλεκτρικά οχήματα, λόγω χάρη. Πρέπει να δούμε τι είναι από βιομηχανική άποψη ρεαλιστικό, από άποψη στρατηγική, τι είναι ένα πιθανό επίπεδο αναγκών σε ηλεκτρισμό για τα οχήματα αυτά, τι υποδομέ χρειάζονται, ποιε θα ήταν οι επιπτώσει για τον ηλεκτρισμό, την ηλεκτρική ενέργεια χωρί άνθρακα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε δηλαδή πολύ περισσότερα οχήματα ηλεκτρικά μεν, αλλά τα οποία να παράγονται από λιθάνθρακα λόγω χάρη, να χρειάζονται εργοστάσια λιθάνθρακα για να παραχθούν. Δεν θα μας ωφελούσε αυτό σε τίποτα. Για τα ραδιενεργά απόβλητα και το χρονοδιάγραμμα για την οδηγία. Με συγχωρείτε, δεν θυμόμαι την ακριβή ημερομηνία. Αλλά νομίζω ότι είχαμε μιλήσει για αναθεώρηση με προπτική πενταετίας και δεκαετίας σε σχέση με τα τώρα προτινόμενα. Οπότε η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ και θα αναθεωρηθεί ε, για, με έναν ε, μακρύ ορίζοντα. Θεωρώ ότι είναι σημαντική συμβολή μια τέτοια στρατηγική ώστε να αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή πυρηνική πολιτική και ενέργεια μπορεί να είναι ασφαλέστερη παγκοσμίω. Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε μια περίοδο αναθεώρησης πιο βραχία και αν χρειαστεί θα το πράξουμε. Τώρα, για, το, για να επανέλθω στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια από, ένας από τους τομείς τους πλέον ενδιαφέροντες, τους πιο συναρπαστικούς που έχουμε στην γενική μας διεύθυνση. Υπάρχει τόσο δυναμικό εδώ. Όμως η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν αφορά το χάσμα, την απόσταση δηλαδή, της προμήθειας που τώρα έχουμε και το τι ζήτηση μπορεί να υπάρχει και της ανάγκης εξοικονόμησης. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όσα παρέχονται, όσα μπορεί κανείς να προμηθεύσει, είναι όπως είπατε και ο κύριος Ζαντό σωστά είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιήσουμε ρεαλιστικά στοιχεία για την ενέργεια. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε εδώ ότι όσο περισσότεροι περιορισμοί για την ενεργειακή αποδοτικότητα υπάρχουν, τόσο πιο εύκολα να χαράξουμε και εμεί την πολιτική μας. Εάν βρούμε ένα τρόπο το περιοριστικό στοιχείο να το ενσωματώσουμε, ώστε και να προγραμματίσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, αυτό θα ήταν πολύτιμο. Αυτό είναι ένα επιχείρημα υπέρ των υποχρεωτικών στόχων άλλωστε. Αλλά όσο και αν μπορώ αυτό να το βεβαιώσω, δεν είμαι σε θέση σήμερα να λάβω μια θέση οριστική για το θέμα. Πάντω σίγουρα το δυναμικό που υπάρχει εδώ δεν το έχουμε αξιοποιήσει πλήρως. Θα πρέπει οι δικέ μας πρακτικές στην Ευρώπη να φτάσουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Και τα δίκτυα, αλλά και τα μέτρα ενεργικής αποδοτικότητας για τις εταιρείε, τα κτίρια και τα νοικοκυριά. Όλα αυτά είναι ένα πεδίο όπου έχουν δοθεί πολλά κονδύλια για ερευνητικά προγράμματα και τεχνολογικά μέσα, αλλά ακόμη δεν έχουμε λάβει αποφάσεις. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρχίζουν να κερδίζουν από αυτά. Και αυτό είναι καλό. Να μπορεί κανείς να βγάζει κέρδος από νέες πρωτοβουλίες. Αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει και το απαραίτητο πλαίσιο για να εργαστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να πετύχει αυτή η προσπάθεια. Δεν ήξερα ότι έχουμε αποδυναμώσει τους στόχους μας και ότι είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις επιδόσεις μας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να το ξαναδώ. Θα ξαναμελετήσω. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι ναι, αυτός είναι ένας από τους πυλώνες της ενεργειακής μας πολιτικής, η ενεργειακή αποδοτικότητα. Σίγουρα υπάρχουν ε, στοιχεία της διαχείρισης και επιπτώσεις που μπορεί να συνηγορούν ε, θερμά υπέρ των ε, υποχρεωτικών στόχων, όμως θα πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά η ισορροπία και η εξίσωση προσφορά και ζήτηση. Ακούσαμε νωρίτερα πολλού να αναφέρουν σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου τέτοια σχόλια που δείχνουν ότι όσοι εργάζονται για την ενέργεια ή το περιβάλλον δεν χαίρονται πολύ που κάποιοι λένε ότι τα ορυκτά καύσιμα παράγουν λιγότερο άνθρακα από άλλα και γι' αυτό είναι καλά, ο στόχος μας είναι να έχουμε μια κοινωνία τελείως απαλλαγμένη από τον άνθρακα ή έστω χαμηλής παραγωγής άνθρακα. Ελπίζω λοιπόν εδώ πραγματικά να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε με όσους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν τον τομέα, ώστε να έχουμε μια λεπτομερή συζήτηση και να δούμε ακριβώς και σε ποιο επίπεδο θα μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Ευρωπαϊκό ή εθνικό ή τοπικό. Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι δεν κάλυψα όλε τι ερωτήσει, αλλά νομίζω ότι σα έδωσα μια πρόγευση για το είδο προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε σε μια σειρά από ζητήματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά που είπατε εσεί και για τι ερωτήσει και τι απαντήσει. Ε, κύριε Γενική Διευθυντά, εγώ βρήκα ιδιαίτερα συμπαθητικό αυτό που είπατε, ότι καλύτερα να προετοιμάζει κανείς ε, τα πράγματα με σωστό τρόπο ε, και να τα φέρνει προς ψήφιση αντί βεβαιεσμένα να θέλει να τα προχωρήσει πάση θυσία. Νομίζω όλοι έχουμε κάνει εμπειρία για αυτόν τον τρόπο εργασίας και νομίζω καλύτερα να παίρνει κανείς το χρόνο του και να δουλεύει αποτελεσματικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στις 3 ε, η ώρα το απόγευμα. Γεια σας.